Κυρίε Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας παρακαλώ καθίστε. Ας αρχίσουμε τη δεύτερη αυτή συνεδρία της διακοινοβουλευτικής μας συνάντησης για την επανεξέταση της στρατηγικής 2020 και προτεραιότητες του 2015 και του κύκλου των Ευρωπαϊκών Εξαμήνων πριν να προχωρήσουμε σε αυτό το θέμα. Να συνοψίσουμε τα σημαντικότερα πορίσματα των τριών επιτροπών, Econ, Empl και Budget, για τα διάφορα θέματα. Η Επιτροπή Οικονομικών συζήτησε δύο θέματα, τον συντονισμό για φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή και την ευθύνη των εποπτικών αρχών για τα τραπεζικά και ιδίως μέσα στην Τραπεζική Ένωση θέματα που είναι απολύτως κρίσιμα και όπου η συνεργασία, θα έλεγα εγώ, μεταξύ των εθνικών και Ευρωπαίων βουλευτών είναι πραγματικά αναγκαία. Για το πρώτο θέμα συζητήσαμε αφενός τα προβλήματα φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής, από την άλλη μεριά τον επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό, φοροαποφυγή και ακούσαμε από τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πώς σκέπτεται να αντιμετωπίσει στο ευρωπαϊκό επίπεδο η Επιτροπή το θέμα αυτό. Οι διάφοροι που έλαβαν το λόγο συμφώνησαν ότι πρέπει να γίνει διάκριση μεταξύ φοροαποφυγής, φοροδιαφυγής και των φοροδιαφυγών που είναι τεχνικά μεν ε, νόμιμοι αλλά είναι και δύσκολο να αντιμετωπιστεί. Πρέπει λοιπόν να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα αυτά. Εγώ νομίζω ότι η αναγνώριση ήταν ομόφωνη ότι πρέπει να αλλάξει το status quo, το, status και ορισμένοι συνάδελφοι ε, κατέθεσαν και συγκεκριμένα παραδείγματα για κάποιες μορφές συνεργασίας. 28 ισπανικές εταιρείες, είπε για παράδειγμα ο κύριος Λάγκεν, μετέφεραν την έδρα τους σε άλλη χώρα και πληρώνουν τους φόρους τους εκεί. Τίθεται λοιπόν το θέμα του ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να πληρώνουν φόρους εκεί όπου ε, γίνεται η παραγωγή του προϊόντος τους, η παραγωγή δηλαδή του πλούτου. Μιλήσαμε και για το διαφορετικό επίπεδο αρμοδιοτήτων και ευθύνης στον φορολογικό χώρο και η διάκριση αρμοδιοτήτων μεταξύ των θεσμικών οργάνων και αυτή βέβαια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι κάπως περιορισμένη. Από την άλλη μεριά τα εθνικά κοινοβούλια έχουν κρίσιμο ρόλο να παίξουν. Συζητήσαμε διάφορες προσεγγίσεις εναρμόνισης, σύγκρισης, συνεργασίας και υπήρξε και ένα κοινό αίσθημα επίγοντος θα έλεγα για το γεγονός ότι χρειάζεται πράγματι να προχωρήσουμε. Καλωσορίζουμε τα πρώτα βήματα που έγιναν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από χώρες μέλη σε διάφορους τομείς, αλλά νομίζω ότι πρόκειται για μια κοινή δέσμευση, δηλαδή να κάνουμε την προσπάθεια και για του χρόνου να επιτύχουμε νέα πράγματα. Γνωρίζετε και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα αρχίσει η σχετική πρωτοβουλία, θα δούμε με ποια νομική μορφή, αν θα είναι εξεταστική επιτροπή, έκθεση, η σχετική απόφαση θα ληφθεί περί τα τέλη της εβδομάδος. Πάντως, με κάθε τρόπο η Ευρωβουλή θα προχωρήσει και σε νομοθετικού χαρακτήρα πρωτοβουλία για το θέμα αυτό και πιστεύω ότι πρέπει να συνεργαστούμε με τα Εθνικά Κοινοβούλια για την σύνταξη αυτής της εκθέσεως. Τώρα για το δεύτερο θέμα αναγνωρίζουμε κάτι που θεωρήθηκε επαναστατικό, δηλαδή η Τραπεζική Ένωση και η εποπτεία στο ευρωπαϊκό τουλάχιστον επίπεδο όλων των τραπεζών και βεβαίως πρέπει να θεσπίσουμε και την accountability. Οι διάφοροι αγορητές μίλησαν για διάφορες νομικές ρυθμίσεις για την εξασφάλιση του ελέγχου και από τα Εθνικά και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και συζητήσαμε επίσης πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την συνεργασία στο εγχείρημα αυτό διότι είναι αναγκαία η ανεξαρτησία, απαιτεί όμως και ένα επίπεδο εποπτείας και λογοδοσίας, accountability δηλαδή. Με την ευκαιρία συζητήσαμε και άλλα στοιχεία που έχουν σχέση με την Τραπεζική Ένωση και την χρηματοδοτική, χρηματοπιστωτική μάλλον ρύθμιση. Είναι ο τρίτος πυλώνας που προσφέρει τις εγγύσεις αυτές όπως είπε η Ρίζα Φερέιρα και μιλήσαμε και για, τις, για την εμπλοκή αυτού του νέου συστήματος εποπτείας και για όλους τους μηχανισμούς εξυγίανσης τραπεζών, αντιμετώπισης κρίσεων, όπου βεβαίως όλοι και όλες ελπίζουμε ότι ο κύριος στόχος θα είναι, που είναι μάλλον, να αποφύγουμε την ανάληψη των βαρών από τους φορολογουμένους σε περίπτωση παρεμβάσεων, σε περίπτωση παγκοσμίων κρίσεων. Και ορισμένοι οι εθνικοί βουλευτές υπενθύμησαν ορισμένα στοιχεία που ελείπουν από το οικοδόμημα αυτό και εμείς τους εξηγήσαμε ποια δουλειά κάνουμε πάνω στον κανονισμό για την διάρθρωση των τραπεζών που είναι ένα νομικό κείμενο το οποίο βρίσκεται υπό συζήτηση τώρα. Αυτά λοιπόν με συνοπτικό τρόπο τα όσα συζητήσαμε. Τώρα ευχαρίστως να δώσω τον ε, λόγο στην Μαρίτα Ουλφσκογκ, πρόεδρο της Επιτροπής Απασχολήσεως. Ευχαριστώ πολύ. Η Διεκνοητική Επιτροπή, η οποία συνήλθε, ασχολήθηκε με δύο συνεδρίες. Η πρώτη αφορούσε την απασχόληση και τους ε, κοινωνικούς δείχτες, δηλαδή το βαθμολόγιο μέσα στα πλαίσια των μακροοικονομικών ανισορροπιών και το δεύτερο αφορούσε το επενδυτικό πρόγραμμα. Πολλοί ομιλητές τόνισαν τη σημασία δημιουργίας απασχόλησης εστιάζοντας την προσοχή σε αξιοπρεπή και στην αξιοπρεπή και ποιοτική εργασία. Το μέλλον μας δεν ε, βασίζεται στην ασταθή εργασία ε, με χαμηλό μισθολόγιο και περιορισμένες δεξιότητες, όπως είπαν πολλοί ομιλητές. Η κυρία Μαρτίνες μίλησε εξ ονόματος της ε, Γερουσίας μίλησε για την φορολογική ολοκλήρωση και εξυγίανση και μίλησε για το γεγονός ότι η ανάπτυξη και η απασχόληση παρουσιάζουν μια θετική εικόνα στην Ισπανία με βάση τις ε, διαρθρωτικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις που έλαβαν χώρα στην Ισπανία τη Σύνοδο Αποκρίσεων και οι εθνικοί βουλευτές και επίσης οι εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μίλησαν για την έλλειψη κοινωνικής ασφάλισης και για το μηδενικό παράγοντα μισθολογίου Επίσης έγινε λόγος για την ανάγκη ενίσχυσης της κοινωνικής διάστασης της ΟΝΕ και την ανάγκη να εισαγάγουμε πιο δυναμικά στοιχεία στην πολιτική μας έτσι ώστε να εντάξουμε και τους αυτόματους μηχανισμούς για τη διόρθωση σφαλμάτων, ιδιαίτερα στον τομέα της ε, φορολογικής και δημοσιονομικής πολιτικής. Το βαθμολόγιο θα πρέπει να σχετίζεται με μια στοχοθέτηση για την ποιότητα εργασίας, κάτι το οποίο έθιξαν πολλοί ευρωβουλευτές και επίσης ότι τα κοινωνικά θέματα και τα θέματα ε, κοινωνικής ενίσχυσης θα πρέπει να τεθούν σε ένα ισόβαθμο πλαίσιο. Ως προς τις επενδύσεις, το σχέδιο ε, επενδύσεων, ο πρόεδρος ε, της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Πολωνικής Γερουσίας μίλησε για την πολιτική θέληση που θα πρέπει να υπάρχει για να επιτύχει το σχέδιο επενδύσεων. Ο κύριος Ντομινίκ Χάνικεν από την Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Ιρλανδικής, του Ιρλανδικού Κοινοβουλίου μίλησε για την ανησυχία του ε, φορολογικού πολλαπλασιαστή καθώς ε, και την εμπράγματη εφαρμογή της ΟΝΕ μέλος της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Απασχόλησης, με συγχωρείτε, τόνισε ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να συνεισφέρουν πολύ περισσότερο στην προσέλκυση εθνικών επενδυτών και ιδιαίτερα τραπεζών για να φτάσουμε στην επίτευξη του πολλαπλασιαστικού παράγοντα. Μπορούμε να πούμε ότι και τα Εθνικά Κοινοβούλια και οι εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού ασχολήθηκαν και τόνισαν την ανάγκη προώθησης των επενδύσεων που θα πρέπει να αποκλειστούν από τον υπολογισμό των εθνικών ελλημάτων σύμφωνα με το πρόγραμμα Juncker και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη το, τη δυναμική της δημιουργίας νέων θέσεων απασχόλησης και τόνισαν και το ρόλο των ΜΜΕ και τη σημασία της επιλογής ενός ευρωπαϊκού τρόπου, όχι αμερικανικού, για να καταβάλουμε προσπάθειες για δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας. που έχουν σημασία για εμάς και για την κοινωνία μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Μαρίτα. Ο Ζαν Αρτούι έχει το λόγο για να μας μιλήσει για τη συζήτηση στην Επιτροπή Προϋπολογισμών. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρόεδρε, το θέμα που επιλέξαμε για την διάσκεψη αυτή της διακοινοβουλευτικής μας συνεδριάσεως ήταν οι οφειλές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καλέσαμε τρεις τοπικούς παράγοντες από την Ισπανία, την Πολωνία και τη Γαλλία να έρθουν να μας παρουσιάσουν αυτά που ζουν επί τόπου εξαιτίας των απλήρωτων λογαριασμών των οφειλών μας και μας εξήγησαν σε τι βαθμό πλήττονται οι επενδύσεις γιατί το βασικό του προπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να στηρίζει τις επενδύσεις. Υπογράμμισαν λοιπόν σε τι βαθμό οι καθυστερημένες πληρωμές δυσκολεύουν τους δικαιούχους των ευρωπαϊκών κονδυλίων και τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις, τα ερευνητικά κέντρα, τους συλλόγου να εκπληρώσουν το έργο τους. Μας εξήγησαν επίσης πώς οι καθυστερήσεις αυτές πλήττουν τους θεμελιώδες μας στόχους, που είναι η ανάπτυξη και η απασχόληση. Επιπλέον, πλήττεται η εμπιστοσύνη των πολιτών και των επενδυτών στην Ευρώπη. Μπορούμε να πούμε ότι όλα αυτά ενισχύουν την κακή εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αν έπρεπε να βγάλουμε μια φωτογραφία για να διαπιστώσουμε την αλλαγή στην εικόνα αυτή, ε, νομίζω ότι τα αποτελέσματα των εκλογών του Μαΐου τα λένε όλα από μόνα τους. Και επιπλέον, γίνεται έλεγχος πολύ γραφειοκρατικός και κατακαιρματισμένος όσον αφορά τις πληρωμές αυτές καθ' αυτές, κάτι το οποίο οδηγεί σε καθυστερήσεις και δυσκολίες. Επιπλέον διαπιστώνουμε δύσκολες σχέσεις ανάμεσα στα Εθνικά Κοινοβούλια και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τα Εθνικά Κοινοβούλια σπάνια ελέγχουν την κυβερνητική πτυχή του ελέγχου του Ευρωπαϊκού Προπολογισμού. Γι' αυτό και ζητήσαμε από τους συναδέλφους μας στα Εθνικά Κοινοβούλια να υπογραμμίσουν στις κυβερνήσεις τους ότι οφείλουν να αναλάβουν πλήρως τις υποχρεώσεις τους. Οι οφειλές ουσιαστικά είναι τα χρέη των χωρών μελών. Και πρέπει να αποφεληθούμε από την ευκαιρία που έχουμε για την αναθεώρηση του πολιτούς δημοσιονομικού πλαισίου, που γίνεται στα μέσα της περίοδου, μια που υιοθετήθηκε πριν καν ανανεωθεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η αναθεώρηση αυτή πρέπει να γίνει και πρέπει να υποφεληθούν από αυτή για να σταματήσουν πια αυτοί οι απλήρωτοι λογαριασμοί που ήταν 5 δισεκατομμύρια το 2010 και που σιγά σιγά έφτασαν στα 25 με 30 δισεκατομμύρια το 2014. Συνεπώς πρέπει να υποχρεώσουμε τις κυβερνήσεις να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Η πολιτική απόφαση είναι μια τέτοια δέσμευση, να γίνονται πληρωμές τότε που πρέπει, γιατί αυτές είναι υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει οι κυβερνήσεις. Πώς να αποφεληθούμε, α, μάλλον να απαλλαγούμε από τις οφειλές αυτές στο μέλλον, προτείναμε την μείωση των προγραμμάτων και είπαμε να φροντίσουν να έχουν πραγματική προστιθέμενη αξία όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα, την ανάπτυξη και την απασχόληση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αποφασίσει ποιες είναι οι προτεραιότητές της και να αποφύγει τον κατακαιρματισμό των πόρων. Πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρξει ευελιξία και πρέπει να αναρωτηθούμε επίσης για το κατά πόσο είναι σωστό να είναι επταετές το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Πιστεύουμε ότι δεν μπορεί να προσαρμοστεί στη συγκυρία κάθε φορά ένα τέτοιο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Οι έλεγχοι μερικές φορές είναι τόσο πολυπληθείς και τόσο κατακαιρματισμένοι που δεν είναι αποτελεσματικοί. Πρέπει να απλοποιήσουμε λοιπόν την αλυσίδα, την ελεγκτική. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αλήθεια και αυτή φταίει μερικές φορές για τους υπερβολικούς ελέγχους αλλά από την άλλη μεριά είναι και οι εθνικές δικήσεις, οι κυβερνήσεις που προσθέτουν και αυτές παραπάνω γραφειοκρατία. Η λύση μεσοπρόθεσμα φαίνεται ότι είναι ένα πραγματικό σύστημα ιδίων πόρων. Αν λοιπόν περιμένουμε προτάσεις από τον κύριο Μόντι και την ομάδα του, αυτό θα μπορούσε να βοηθήσει. Σήμερα το απόγευμα συζητάμε για την αναθεώρηση της στρατηγικής ε, ενόψης του 2020 και το ευρωπαϊκό εξάμεινο. Σίγουρα οι επενδύσεις μπορούν να βοηθήσουν πάρα πολύ τους στόχους στρατηγικής 2020 και τις προτεραιότητες που αναφέρονται στο ευρωπαϊκό εξάμεινο. Έχουμε πάρα πολλούς κανόνες, αλλά ελάχιστα εργαλεία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το θέμα των οφειλών πρέπει οπωσδήποτε να τακτοποιηθεί ώστε ο προπολογισμό μας να μπορεί να φέρει σε πέρας τους στόχους μας. Δεν πρέπει να υπάρχει επιφυλεκτικότητα. Η Ευρώπη μπορεί να προχωρήσει μόνο εφόσον έχει την εμπιστοσύνη των πολιτών και εμπιστοσύνη δεν μπορεί να υπάρχει όταν παραμένουν οφειλέ. Για να πετύχει το επενδυτικό σχέδιο των 315 δισεκατομμυρίων πρέπει να υπάρχει εμπιστοσύνη και από πλευρά ε, των πολιτών και από πλευρά των επενδυτών οφείλουμε να τηρήσουμε τις υποχρεώσεις μας, χωρίς καθυστερήσεις. Σας ευχαριστώ αγαπητέ συνάδελφε και τώρα μπορούμε να αρχίσουμε την πραγματική μας συνεδρίαση Ολομέλειας ε, για την αναθεώρηση στρατηγικής 2020 και για τις προτεραιότητες του κύκλου των Ευρωπαϊκών Εξαμήνων 2015. Πρώτα θα ήθελα να απευθύνω το καλώς ορίσατε στον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμόδιο για απασχόληση και ανταγωνιστικότητα κύριο Κατάινεν. Καλώς ήρθατε αγαπητέ κύριε Επίτροπε στη διακοινοβουλευτική μας συνάντηση και λαμβάνετε αμέσως το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Γκουαλτιέρη σας ευχαριστώ. Είναι τιμή για μένα και ευχαρίστηση που με προσκαλείτε στη σημαντική αυτή διακοινοβουλευτική εβδομάδα για να συζητήσω μαζί σας σημαντικά θέματα τη στρατηγική δηλαδή της Ευρώπης 2020 και το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο 2015. Δυστυχώς και οφείλω να σας ζητήσω συγγνώμη για την ανάγκη να εγκαταλείψω την αίθουσα ε, τι έχω αντιλημμένες υποχρεώσεις, αντιλημμένες υποχρεώσεις αργότερα. Βεβαίως θα συνεχίσουμε τον διάλογο. Από τη δική μου πλευρά οφείλω να πω ότι χαίρομαι πολύ που βλέπω τόσους πολλούς εθνικούς βουλευτές παρόντες εδώ και παρούσες βεβαίως. Το 2010 εγκρίθηκε η Ευρώπη 2020 ως μακροπρόθεσμο όραμα για το κοινωνικό και οικονομικό πρότυπο. Μετά από αυτά τα πρώτα χρόνια, το πρώτο μισό δηλαδή, της εφαρμογής της, είναι χρήσιμο να σταματήσουμε να προβληματιστούμε. Αυτό είναι και ο στόχος της επανεξέτασης της στρατηγικής που αναλαμβάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η πρόοδος προς την επίτευξη των στόχων είναι άνηση, πολύ άνηση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται αρκετά κοντά στην ορθή πορεία για θέματα όπως παιδεία, κλίμα και ενέργεια. Δυστυχώς αυτό δεν μπορεί ε, να λεχθεί για άλλους στόχους όπως της απασχόλησης, έρευνα, έρευνας και ανάπτυξης και μείωσης της φτώχειας. Η οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση στην Ευρώπη βεβαίως είχε σημαντικά θύματα. Οι χώρες μέλη δεν μεταρρύθμισαν σημαντικούς τομείς των οικονομιών τους και υπολείπονται των στόχων τους. Η ανανεωμένη δέσμευση για τους διαρθρωτικούς στόχους για την αύξηση της ανάπτυξης και της απασχόλησης είναι λοιπόν ε, μή κλειδιά για την ανάπτυξη και την απασχόληση. Να πω λίγα λόγια για το πώς προτιθέμεθα να προχωρήσουμε. Τον Μάρτιο του 2014 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση για τη στρατηγική 2020, την πρόοδο που είχε επιτευχθεί μέχρι τότε και το που βρισκόταν η κατάσταση. Μετά από την ανακοίνωση αυτή διεξήχθη δημόσια διαβούλευση για την Ευρώπη 2020 από τις 5 Μαΐου 2014 μέχρι την 1η Οκτωβρίου του ίδιου χρόνου. Με στόχο να συγκεντρωθούν ιδέες όλων εκείνων που εμπλέκονται στην εφαρμογή της στρατηγικής. Έμαθα λοιπόν από την εμπειρία αυτών και τις βέλτιστες πρακτικές τους. Έλαβε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχεδόν 800 συνεισφορές σε αυτή τη δημόσια διαβούλευση. Σύντομα θα υποβάλουμε έγγραφο με τα σχετικά συμπεράσματα. Θα προχωρήσουμε και στην επανεξέταση την άνοιξη του 2015 της στρατηγικής μας για το 2020. Βεβαίως υπάρχουν και άλλες προτεραιότητες και γι' αυτό προτιμούμε να προβληματιστούμε περισσότερο και να αναμένουμε λίγο περισσότερο για να υποβάλουμε τι προτάσει για την επανεξέταση. Έτσι λοιπόν τα επόμενα βήματα θα έχουν ως εξή. Πρώτα ως Κομισιόν θα υποβάλουμε μια περίληψη των βασικών συμπερασμάτων που προκύπτουν από την δημόσια διαβούλευση μαζί με μια έκθεση για το που βρισκόμαστε, state of play δηλαδή, για τους στόχους 2020. Αργότερα η Κομισιόν θα υποβάλει προτάσεις για την επανεξέταση της στρατηγικής. Τους επόμενους μήνες, ή επόμενοι μήνες μάλλον, θα παίξουν κέριο ρόλο για την περιγραφή του ρόλου της Ένωσης για τα επόμενα χρόνια. Έτσι λοιπόν εκδηλώσεις όπως η σημερινή είναι σημαντικές για την ενίσχυση των ε, διαλόγων μεταξύ των θεσμικών οργάνων και των ενδιαφερομένων μερών. Η ΔΕΕ Ευρωβουλή έχει παίξει σημαντικό ρόλο από τότε που ξεκίνησε η εκστρατεία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι αυτή η δέσμευση υπέρ μια στρατηγική ανάπτυξη και απασχόληση θα συνεχιστεί τα επόμενα χρόνια. Επιτρέψτε μου τώρα να έρθω στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο 2015 από τα βασικά εργαλεία εφαρμογής στρατηγική 2020. Η Επίτροπος κυρία Τάισεν θα ασχοληθεί περισσότερο με θέματα του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου όταν θα λάβει αυτή το λόγο. Εγώ λοιπόν θα δώσω περισσότερη έμφαση στην διασύνδεση μεταξύ του εξαμήνου και του σχεδίου επενδύσεων. Εισαγωγικά στις 28 Νοεμβρίου η Επιτροπή υπέβαλε την ε, Annual Growth Survey από τον προηγούμενο χρόνο όπως είπα. Πρώτον, αύξηση των επενδύσεων. Δεύτερον, επιτάχυνση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Και τρίτο, δημοσιονομική εξυγίανση η επιθεώρηση, ε, η επιθεώρηση περιγράφει και τα σχετικά με τις επενδύσεις. Λίγα λόγια. Το σχέδιο επενδύσεων βασίζεται σε ένα τρίγωνο. Πρώτα, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Εσείς τώρα εξετάζετε το σχέδιο κανονισμού και αναμένουμε τη διεξαγωγή διαλόγου μαζί σας για να υλοποιηθεί το συντομότερο δυνατό. Δεύτερο, οι επενδύσεις που βρίσκονται στον αγωγό και ο άξονας τεχνικών συμβουλών. Ταξιδεύοντας σε όλες τις χώρες μέλη, θεωρώ ότι αυτό ε, είναι από τα σημαντικότερα στοιχεία. Αυτοί λοιπόν οι δύο πυλώνες θα επιτρέψουν να ξεκινήσουν ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις, ιδίως σε χώρες που έχουν μεγάλα κενά στις επενδύσεις. Τρίτο, λοιπόν, για την πρωτοβουλία, για την επενδυτική πρωτοβουλία, για να μπορέσει αυτή δηλαδή να έχει διαρκή αποτελέσματα, χρειάζονται διαρθρωτικές αλλαγές που να καλύψουν όλη την ενιαία αγορά. Ακόμα δεν έχει καθοριστεί η συγκεκριμένη ατζέντα, το συγκεκριμένο θεματολόγιο. Γνωρίζουμε όμω ήδη ότι η Ενεργειακή Ένωση και η ψηφιακή ενιαία αγορά θα παίξουν σημαντικό ρόλο σε αυτά και πάλι όταν θελήσουμε ε, να τα μεταφέρουμε αυτά σε συγκεκριμένε συστάσει για το εξάμεινο θα πρέπει να παίξουμε βέβαια και εμεί το ρόλο μα. Ολοκληρώνω λέγοντα ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένει με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τι δικέ σα απόψει της Ευρωβουλή, δηλαδή γνωρίζοντα ότι η Ευρωβουλή έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και για την πολιτική επενδύσεων έχοντα δείξει και σχετικά δείγματα στο παρελθόν. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρο Γκουαλτιέρη. Ευχαριστώ, κύριε Αντιπρόεδρε. Δυστυχώ η κυρία Τάισεν ακόμα δεν ε, έχει προλάβει να φτάσει. Άρα λοιπόν θα αρχίσουμε αμέσως με το δεύτερο βήμα που είναι η λήψη του λόγου από τους εισηγητές πρώτα της Οικονομικής Επιτροπής για το HES. Εμείς βεβαίως, απαντώ στον κύριο Κατάινεν, ε, ασφαλώς και έχουμε δεσμευτεί για να προωθήσουμε ταχύτατα τον κανονισμό. Τώρα προχωρούμε σε συνεννόηση μεταξύ των κοινοβουλευτικών επιτροπών. Ασφαλώς θα φανούμε ενεργητική και θα περιμένουμε βεβαίως και τη δική σας συνεργασία για να συζητήσουμε τον σχεδιασμό αυτό, τον οποίο θα συσχολιάσουμε και αύριο στις εργασίες του αυριανού πρωινού. Πρώτα θα δώσω το λόγο στον κύριο Ροζάτη για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, εισηγητής δηλαδή στην Επιτροπή Οικονομικών. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Επίτροπο Κατάινεν γιατί μας έδωσε μια συνολική εικόνα για το ευρωπαϊκό εξάμεινο και τη σύνδεσή του με τη Στρατηγική Ευρώπη 2020. Ήμουν σκιώδης στο... στην προηγούμενη έκθεση σε σχέση με τις συστάσεις προς συγκεκριμένες χώρες και τώρα είμαι για την συνετήση έκθεση ανάπτυξης. Έτσι μπορούμε να ορίσουμε ποια είναι τα προβλήματα σε αυτή τη διαδικασία συντονισμού πολιτικών. Όπως είπατε, στα πλαίσια της οικονομικής διακυβέρνησης θα πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας στο γεγονός ότι έχουμε να κάνουμε με νέες προκλήσεις από την ε, ε, σχετικά αδύναμη ανάπτυξη και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και την κατάσταση αναχώρα. Παράλληλα, θα πρέπει να κάνουμε χρήση των διδαγμάτων που αποκομίσαμε από τον προηγούμενο κύκλο Δηλαδή δεν ήμασταν και ιδιαίτερα αποτελεσματικοί στις συστάσεις προς ε, συγκεκριμένα κράτη-μέλη. Πιστεύω ότι έχουμε να κάνουμε με μία εφαρμογή των συστάσεων το 2013 και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να καταβάλουν κάθε προσπάθεια για να εφαρμόσουν τις συστάσεις αναχώρα. Και επίσης θα πρέπει να μιλήσουμε σε συγκεκριμένες χώρες για συστάσεις και ζητήματα που θα πρέπει να αντιμετωπίσουν. Επίσης θα πρέπει να υπάρξει κινητοποίηση του πολιτικού αυτού κεφαλαίου μέσα στα πλαίσια των συστάσεων ετήσια έκθεση ανάπτυξης είναι ένα βασικό έγγραφο που σχετίζεται με το συντονισμό των πολιτικών μεταξύ κρατών μελών. Ελπίζω να μπορέσουμε να έχουμε μία προσέγγιση με βάση τα δεδομένα και γνώμονα της συστάσης της Επιτροπής και να λάβουμε υπόψη τις συγκεκριμένες δράσεις για το μέλλον. Πιστεύω όμως ότι υπάρχει συνένεση ότι οι τρεις πυλώνες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποτελούν την κατάλληλη προσέγγιση. Ο πυλώνας των επενδύσεων είναι ύψης της σημασίας για να αντιμετωπίσουμε το έλλειμμα εμπιστοσύνης. Ζούμε έναν φαύλο κύκλο όπου οι χαμηλές επενδύσεις οδηγούν σε χαμηλή ανάπτυξη και η χαμηλή ανάπτυξη σε χαμηλή εμπιστοσύνη η οποία στρέφεται σε χαμηλές επενδύσεις με τη σειρά της. Γι' αυτό θα πρέπει να σπάσουμε αυτό το φαύλο κύκλο και υπ' αυτή την έννοια καλωσορίσουμε την έκθεση AGS της Επιτροπής που θέλει να σπάσει αυτό τον φαύλο κύκλο έχει μεγάλη σημασία ιδιαίτερα στα κράτη-μέλη που έχουν επαρκή δημοσιονομικό πλαίσιο και προσανατολισμούς που έχουν συγκεκριμένα, ένα συγκεκριμένο πάτημα για την οικονομική ανάπτυξη και μπορούν να ευεργετηθούν από το Ταμείο αυτό. Επίσης, θα πρέπει οι αγορές εργασίας να γίνουν πιο αποτελεσματικές για να εξυγχρονίσουμε το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης και το σύστημα συνταξιοδότησης με βάση και τα πλαίσια της γενικότερης σταθερότητας. Θα ήθελα να πω ότι δίνουμε μεγαλύτερη έμφαση στις ΜΜΕ που θα πρέπει να έχουν ε, ευκολότερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση, όχι μόνο από το EFCI, αλλά και από εναλλακτικές πηγές ε, τραπεζικών ε, επενδύσεων, δηλαδή κεφάλαια κινδύνου ή ομότιμα κεφάλαια, κεφάλαια προς ομότυπους, ομότιμους, έτσι ώστε να μπορέσουν να έχουν περισσότερη και καλύτερη πρόσβαση. Επίσης, αυτό που έχει σημασία στη δημοσιονομική εξυγίανση είναι να ανοικοδομήσουμε την εμπιστοσύνη χωρίς να έχουμε βεβαίως υπερβολικά επίπεδα χρέους, γιατί διαφορετικά δεν είναι δυνατόν να οικοδομηθεί εμπιστοσύνη και να υπάρξει ανάπτυξη. Σε σχέση με τον τρίτο πυλώνα, δηλαδή τις ε, διαρθρωτικές ε, μεταρρυθμίσεις μέσα στα πλαίσια της ε, ετήσιας επισκόπησης της ανάπτυξης, αυτό που έχει σημασία είναι να εντάξουμε αυτά τα δεδομένα στη Στρατηγική Ευρώπη 2020. Όταν μιλάμε για ειδικές συστάσεις προς τα κράτη, η Επιτροπή θα γνωστοποιήσει στα κράτη-μέλη ποιες είναι οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που θα πρέπει να εφαρμόσουν για να φτάσουν στους στόχους της Ευρώπης 2020. Οι στόχοι της Ευρώπης 2020 ε, αποτελούν μια πολιτική δέσμευση καθαρά. Δηλαδή όλοι οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα πρέπει να τηρήσουν αυτό το πλαίσιο. Ελπίζω η ενδιάμεση αναθεώρηση της Ευρώπης 2020 από την Επιτροπή θα μας δείξει κατά πόσο προχωρούν οι χώρες, γιατί δεν προχωρούν όλες με τον ίδιο ρυθμό και υπάρχουν καθυστερήσεις οι οποίες δεν θα πρέπει να συνεχιστούν στα κράτη-μέλη. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να επιταχύνουν την όλη διαδικασία. Τέλος, θα ήθελα να πω ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο είναι μία βασική συνιστόσα της οικονομικής ε, διακυβέρνησης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί δεν χρησιμοποιούμε αυτό το μέσο εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα διασφαλίζει τις σωστές ε, διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στα κράτη-μέλη. Το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο ε, δεν είναι τέλειο αυτή τη στιγμή και ολοκληρωμένο, αλλά αποτελεί μια πολύ καλή βάση και θα μπορούσε να είναι και πιο φιλικό. Από τα στοιχεία που λαμβάνουμε από τα κράτη-μέλη, θεωρούμε ότι μπορούμε να έχουμε σκόπιμες ενδείξεις για το πώς θα μπορέσουν να δράσουν και οι εθνικοί παράγοντες. Επίσης, θα πρέπει να ενισχύσουμε το εθνικό πλαίσιο αναφοράς. Πρόκειται για ένα εγχείρημα το οποίο προωθούμε για τα κράτη-μέλη. Δεν είναι κάτι που επιβάλλεται εκ των έξω και δεν θα πρέπει να θεωρηθεί όχληση είναι, πρόκειται για συμβουλές που θα πρέπει να ακολουθήσουν τα κράτη-μέλη, αλλά θα πρέπει και οι κυβερνήσεις και τα εθνικά κοινοβούλια να ιδιοποιηθούν αυτά τα δεδομένα. Γι' αυτό θεωρούμε ότι τα εθνικά κοινοβούλια θα πρέπει να συμμετέχουν πολύ περισσότερο. Ευχαριστούμε πολύ τον ε, Ντάρις Ροσάτη. Ε, θα δώσω το το λόγο στον κύριο Σέρζο Γκουτιέρες Πριέτο από την Επιτροπή Απασχόλησης. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο είναι ένας από τους πιο σημαντικούς συντονιστικούς ε, μηχανισμούς και μάλιστα ο μοναδικός που έχουμε στη διάθεσή μας, αλλά ένας μηχανισμός που έχει χρησιμοποιηθεί στραβά. Γιατί αυτό που λείπει είναι ο συντονισμός των πολιτικών που σχεδιάζονται με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη και αυτό που λείπει κυρίως είναι η συμμετοχή των Εθνικών Κοινοβουλίων σε αυτόν. Δεν υπάρχει δηλαδή δημοκρατική νομιμότητα. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε με αυτή τη διαδικασία, αλλά πιστεύουμε ότι δεν καλύπτεται με την κατάσταση που έχουμε σήμερα. Γιατί από την αρχή, από τη στιγμή δηλαδή που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν καν έχει την έκθεσή της για την ανάπτυξη, αρχίζει διάλογο με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Αυτό όμω τι σημαίνει. Σημαίνει ότι οι χώρες μέλη πρέπει να παρουσιάζουν τα δικά τους τα προγράμματα, αλλά προηγουμένως να έχουν ενημερώσει και να τα έχει εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πολλά λοιπόν μπορούμε να βελτιώσουμε σε αυτή τη διαδικασία, ώστε τα εθνικά κοινοβούλια να νιώσουν μέρος της διαδικασίας και προκειμένου να υπάρχει αυτή η δημοκρατική νομιμότητα και αποτελεσματικότητα. Γιατί αν τους συνομοθέτες από τις χώρες μέλη τους αποκλείουμε από τη διαδικασία, κάνουμε βήματα προς τα πίσω. Αντί να βελτιώνουμε την ανταγωνιστικότητα και τον συντονισμό των οικονομιών μας. Συνεπώς, παρόλο που το βάζει τρίτη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να μπει στην πρώτη θέση η ενίσχυση της δημοκρατικής νομιμότητας και της συμμετοχής των ε, βουλευτών από τα Εθνικά Κοινοβούλια. Τώρα, από εκεί και πέρα, εμείς θέλουμε να έχουμε μια έκθεση για να βελτιώσουμε την οικονομική κατάσταση, η οποία φυσικά είναι βάλωτη, το βλέπουμε κάθε χρόνο. Λίγο πάνω από 0% ήταν η ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν διαπιστώνουμε νέες θέσεις απασχόλησης, το να μειωθεί απειροελάχιστα η ανεργία δεν είναι αυτά τα αποτελέσματα. Και έτσι καλλιώς αυτό γίνεται με άδικο τρόπο. Δεν δηλαδή ενισχύεται η ισότητα, αντίθετα. Η, στην έκθεσή μας λοιπόν στην Επιτροπή Απασχόλησης είναι να βασιστούμε σε τέσσερις πυλώνες. Πρώτον, πόλα. να δούμε τα κίνητρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μια νέα στρατηγική αλλά πρέπει να είναι ακόμα πιο φιλόδοξη στόχη. Εμείς πιστεύουμε ότι είναι ε, σημαντικό να έχουμε αναθεώρηση του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, αλλά πιστεύουμε ότι πρέπει να μειωθεί αυτή η υπερβολική λιτότητα. Πρέπει να υπάρξει λοιπόν αυτή η αναθεώρηση και στα πλαίσια της αναθεώρησης αυτής να είμαστε πιο ευέλικτοι. Να αναρωτηθούμε δηλαδή θα βοηθήσουν όλα αυτά στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Επίσης πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό να αναθεωρήσουμε και όλη τη στρατηγική των διορθωτικών μεταρρυθμίσεων, κυρίως πάλι σε σχέση με την απασχόληση. Γιατί στην προηγούμενη θητεία, η προηγούμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπάθησε όλη τη στρατηγική κατά πρώτο στάδιο να τη βάλει στη λιτότητα και μετά στις μεταρρυθμίσεις, χωρίς όμως να δει τις ε, προκυκλικές ε, με τα, τα, τα προκυκλικά αποτελέσματα που είχαν όλα αυτά. Αυτό έκανε η Επιτροπή Παρόζο. Το αποτέλεσμα ήταν περισσότερες ανισότητες. Συνεπώς, από την πλευρά της Επιτροπής Απασχόλησης λέμε ότι δεν πρέπει να φτιάξουμε ένα μάντρα, δηλαδή σώνει και καλά διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, να δούμε ποιες είναι αυτές που εξυπηρετούν τους στόχους μας. Έχουν προκυκλικό αποτέλεσμα, θα δημιουργήσουν απασχόληση ή θα ενισχύσουν τις ανισότητε Εργασιακή μεταρρύθμιση, για παράδειγμα. Επικεντρώσαμε πάρα πολύ την προσοχή μας στα εργασιακά. Αποτέλεσε ένα παράδειγμα. Είπαμε ότι έτσι θα δημιουργηθούν περισσότερες θέσεις απασχόλησης. Δεν είναι αλήθεια όμω. Υπάρχουν και άλλες πολιτικές, όπως οι επενδύσεις, που μπορούν επίσης να ενισχύσουν την απασχόληση. Υπάρχει μια συνεχής αντίφαση ανάμεσα στους, στους επιτρόπους ανάμεσα σε αυτούς που ασχολούνται με τα οικονομικά και αυτούς που ασχολούνται με την απασχόληση. Και γιατί, γιατί ενώ στην ετήσια επισκόπηση ανάπτυξης ασχολούμαστε πάρα πολύ με τις διαφορετικές μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται, η Επίτροπος για την Απασχόληση είπε ότι αυτή η εργασιακή μεταρρύθμιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είχε δύο αποτελέσματα. Κατακαιρματισμό πρώτα απ' όλα της αγοράς εργασίας μας η ίδια Επιτροπή το λέει στο παράρτημά της για την απασχόληση ότι 51% της απασχόλησης που δημιουργείται έτσι δεν εξυπηρετεί τους Ευρωπαίους πολίτες για να βγουν από τη φτώχεια. 51% δηλαδή από τις νέες θέσεις απασχόλησης που δημιουργούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αμείβονται με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν με αξιοπρέπεια να ζουν από την εργασία τους Ευρωπαίοι πολίτες. Ναι, εργασικέ μεταρρυθμίσει που οδήγησαν σε μείωση των μισθών σε ορισμένε χώρε, κυρίω στη Νότια Ευρώπη, ήταν υπερβολική αυτή η μείωση. Μείωσε την εσωτερική ζήτηση και έδωσε την εντύπωση στους πολίτες ότι με μεγάλη ανισότητα βγαίνουν από αυτή την κρίση. Συνεπώς, το πρόβλημα είναι και μεταξύ των διαφορετικών ε, γενεών. Έχει γίνει κατακαιρματισμός που καταστρέφει και την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών. Πρέπει να επενθυμίσουμε ότι η απασχόληση είναι κάτι παραπάνω από ένα δικαίωμα. Είναι ομφάλιος, ομφάλιος ε, λόρος για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τα προβλήματα κοινωνία. Κάτι άλλο που αναφέρουμε στην έκθεσή μας είναι η βελτίωση του κοινωνικού μεντέλου μοντέλου που επιδεινώθηκε τον τελευταίο καιρό με την οικονομική κρίση ως αποτέλεσμα των περιβολικών πολιτικών λιτότητας. Για να μειωθούν οι ανισότητες λοιπόν, για να αντιμετωπιστεί αυτό το νέο κύμα ένδυας που δημιουργείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και για να αντιμετωπιστεί ο ευρωσκεπτικισμός και ο λαϊκισμός που είναι επίσης μεγάλα προβλήματα που χτυπάνε σήμερα το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα αυτά πιστεύουμε ότι ναι, δεν μπορούμε να γνωρίσουμε ότι έχει υπάρξει μια σημαντική αλλαγή στην ευρωπαϊκή πολιτική τους τελευταίους μήνες. Αλλά αναρωτιόμαστε, οι αλλαγές αυτές θα εξυπηρετήσουν, θα βοηθήσουν για να βγούμε με φερεγγιότητα και γρήγορα από την οικονομική κρίση. Γιατί η προσωπική μου εντύπωση είναι ότι η Επιτροπή Γιουνκέρ έκανε ό,τι μπορεί προκειμένου η ευρωπαϊκή οικονομία να μην νιώσει την ύφεση, αλλά δεν έκανε ό,τι μπορούσε για να βγούμε από την κρίση. Εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να στηρίξουμε πιο φιλόδοξες ακόμα αλλαγές. Το επενδυτικό σχέδιο, πέρα των σχολείων που κάνουμε κατά πόσο θα είναι αρκετά, κατά πόσο θα αποδώσουν όπως θα θέλαμε, πιστεύουμε ότι πρέπει να αναλάβουν και κινδύνους. Οι επενδύσεις δεν μπορούν να αντικαταστήσουν επενδύσεις που έτσι καλώς θα γινόντουσαν. Και κυρίως να πάνε εκεί που χρειάζονται περισσότερο. Το σχέδιο Juncker δηλαδή πρέπει να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά υπέρ της ανάπτυξης και της απασχόλησης. Μας απασχολεί κυρίως το να μην αντικαταστήσει χρήματα που έτσι καλώς θα επενδύονταν. Όπως είπε και συγκητής από την Οικονομική Επιτροπή, χρειάζεται πιο μεγάλη στήριξη στι μικρέ και μεσαίε επιχειρήσει για να έχουν πρόσβαση σε πιστώσει. Και χρειάζεται να γίνει συζήτηση για την αναδιάρθρωση του ιδιωτικού χρέου. Εμεί δεν την προσέχουμε αρκετά, αλλά αυτή είναι υπεύθυνη για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες στη συνέχεια μπορούν να δημιουργήσουν απασχόληση. Και απασχόληση πρέπει να είναι ποιότητα με καλούς μισθούς, που να ενισχύουν την ανάπτυξη. Πρέπει επίσης να αρχίσουμε τη συζήτηση, η οποία έγινε λιγάκι και όταν ανέλαβε καθήκοντα η Επιτροπή Γιούγκερ, και αυτό είναι η δυνατότητα ενός ευρωπαϊκού πλαισίου ελάχιστων μισθών, για να σταματήσει αυτό το φαινόμενο της εργασιακής ένδυας. Πιστεύουμε ότι υπάρχουν προβλήματα με τις προσωρινές συμβάσεις, περιορισμένου χρόνου δηλαδή, υπάρχουν αυτοί που θέλουν να δουλεύουν πλήρη απασχόληση και που δεν τα καταφέρνουν. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να δούμε η απασχόληση να είναι τέτοια που να προσφέρει αξιοπρεπή ζωή, να συνάδει με την προστασία του περιβάλλοντος κλπ. κλπ. Να δούμε δηλαδή ποια πρέπει να είναι τα χαρακτηριστικά της εργασίας υπενθυμίζουμε ότι και η κοινωνική διάσταση πρέπει να επανεισαχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Την έχουμε βάλει στο πλάι. Συζητάμε για την Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Ναι, αλλά αν η αναθεώρησή της έχει σαν αποτέλεσμα να χάσουμε την κοινωνική διάσταση, εμείς δεν θα συμφωνήσουμε. Υπάρχει μια αλλαγή λοιπόν στην τάση που πρέπει να ενισχυθεί και πρέπει να φροντίσουμε να είμαστε πιο φιλόδοξοι για να ενισχύσουμε την ανάπτυξη και να την νιώσουν όλοι οι πολίτες. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Τώρα θα δώσω το λόγο στον Ανδρέα Σφαμπ που θα μας παρουσιάσει την ε, έκθεση της ε, διακυβέρνησης νέας αγοράς από την Επιτροπή ΙΝΚΟ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι συνάδελφοι. Η συζήτηση για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο περιλαμβάνει και γενικότερους ε, πολιτικούς προβληματισμούς. Τώρα, μία παράμετρος της ανάπτυξης αλλά και του κοινοβουλευτικού ελέγχου που θα μπορούν να ασκούν Εθνικές Βουλές και Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στα πλαίσια της συναπόφασης είναι και ο τρόπος πώς ε, εξελίσσεται η διακυβέρνηση της ενιαίας αγοράς. Χαίρομαι που ο κύριος Γκουτιέρες με την ομιλία του μου πρόσφερε βάσεις για να συνεχίσω εγώ, με την έννοια δηλαδή ότι οι χώρες μέλη λαμβάνουν τα κείμενα του ε, Συμβουλίου των Υπουργών, τα οποία ΣΥΝΑ αποφασίζει. Αυτά λοιπόν τα νομοθετήματα οφείλουν να εφαρμοστούν αποτελεσματικά στις χώρες μέλη με τέτοιον τρόπο ώστε να υποφεληθεί πραγματικά τελικά η ενιαία αγορά. Σύμφωνα με μελέτες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εφόσον συμβεί αυτό, μπορούμε να παραγάγουμε 2% παραπάνω ανάπτυξη χωρίς κανένα άλλο μέτρο περιοριστικό ή διαφορετικό στις ε, χώρες μέλη. Όταν ακούω τώρα τους διάφορους προβληματισμούς που προβάλλονται στο ε, Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και που καμιά φορά με βρίσκουν σύμφωνο συχνά όμως όχι, από τη σκοπιά του Ευρωπαίου νομοθέτη βρίσκω ότι είναι εκπληκτικό το γεγονός ότι διαθέτουμε αυτές τις δυνατότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ωστόσο δεν τις έχουμε εκμεταλλευτεί και πάντως όχι σε επαρκή βαθμό. Γι' αυτό κύριε Πρόεδρε, εξ και της κυρίας Γκαλπέσης ηγητρίας μας που σήμερα κολλείεται, τονίζω ότι η ενιαία αγορά από τη δική μας σκοπιά αποτελεί σημαντικότερο θεμέλιο λίθο, θα πρέπει να παίξει σημαντικότερο ρόλο στα πλαίσια του ε, Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, γιατί από αυτά μπορούμε να δούμε εάν οι χώρες μέλη, είτε πρόκειται για του Βορρά, του Νότου, της Ανατολής ή της Δύσεως, πραγματικά εφαρμόζουν την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία με τον στόχο να καταστήσουν αποτελεσματική την ενιαία αγορά υπέρ των πολιτών η εξέταση της ενιαίας διακυβέρνησης εντός του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου γίνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εμείς υποστηρίζουμε ως Επιτροπή Ενιαίας Αγοράς αυτή την προσπάθεια. Ελπίζουμε ότι θα καταστεί δυνατό σε συνεργασία με τις Εθνικές Βουλές να αποδείξουμε ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο δεν είναι απλά ένας πειραματισμός αλλά ότι στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου οφείλουμε να θέσουμε και συγκεκριμένα θέματα. Γιατί ορισμένες χώρες μέλη δεν εφαρμόζουν όπως πρέπει τις ρυθμίσεις της ενιαίας αγοράς, αφού εν τέλει μπορεί με τον τρόπο αυτό να παραχθεί ανάπτυξη χωρίς επιπρόσθετη επιβάρυνση. Σε αυτά μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο λοιπόν η έκθεση περί ενίας αγοράς και ελπίζω αυτό να συζητηθεί ακόμη περισσότερο και με τις χώρες μέλη. Thank you. Now we can Ευχαριστώ. Τώρα μπορούμε να δώσουμε το λόγο για την συζήτηση. Ήδη έχω λάβει 11 αιτήσει λήψεως λόγου. Έχουμε όμως χρόνο. Μπορείτε αν θέλετε και άλλοι να ζητήσετε να λάβετε το λόγο. Σας παρακαλώ στείλτε μας ε, το έντυπο καταχωρήσεως. Πρώτος ο μιλητής Μανουέλ Σάραζιν από τη γερμανική Bundestag. Κυρίες και κύριοι, το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο είναι από τα σημαντικότερα εργαλεία για την επίτευξη των στόχων Ευρώπης 2020 και σε τομείς όπου οι χώρες μέλη έχουν αποκλειστική αρμοδιότητα ή όπου υπάρχει ε, συντρέχουσα αρμοδιότητα με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο σήμερα δεν καλύπτει επαρκώς ορισμένους τομείς. Η δημόσια συζήτηση περί του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου δεν γίνεται με επαρκή τρόπο. Το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο δεν έχει λάβει αρκετά πολιτικό χαρακτήρα. Η συζήτηση που διεξάγεται γύρω από αυτό είναι τεχνοκρατική και διέπεται κυρίως από τις τοποθετήσεις της Κομισιόν και των κυβερνήσεων. Τα ευρωπαϊκά επιχειρήματα δεν βρίσκουν απήχηση στις συζητήσεις που γίνονται στις χώρες μέλη, συζητήσεις οι οποίες διεξάγονται εν τέλει σαν να πρέπει οι χώρες μέλη να αμήνονται απέναντι στις Βρυξέλλες. Ούτε οι στόχοι της Ευρώπης 2020 συζητούνται για το πώς θα εφαρμοστούν δεσμευτικά στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξάμεινου. Μπορεί λοιπόν να βελτιωθεί το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο με καλύτερη συμμετοχή των εθνικών βουλών. Εδώ νομίζω ότι πρέπει να κάνει κανείς ορισμένες προτάσεις. Και πρώτο, η ετήσια επισκόπηση ανάπτυξης στο μέλλον να συζητείται σε διαδικασία συναποφάσεως μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Η ευρωπαϊκή συζήτηση λοιπόν να ενισχυθεί. Από την άλλη μεριά θα ήθελα να ενισχυθούν οι εθνικές βουλές και τα εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων μετά από τις συζητήσεις στις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές τους και στις Ολομέλειες. Έρχονται τελικώς τα θέματα αυτά στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Νομίζω όμω ότι οι εθνικέ βουλέ πρέπει να βρίσκονται και σε διαρκή επαφή με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και μάλιστα όχι μόνο για να προβάλλουν εθνικά επιχειρήματα απέναντι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και για να δοθεί η δυνατότητα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενδεχομένω και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να μπορούν να υποβάλουν τα δικά του επιχειρήματα στι εθνικέ κοινέ γνώμε. Γι' αυτό προτείνω σε κάθε, Ευρωπα... σε κάθε Εθνική Βουλή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έρχεται να παρουσιάζει το σχέδιο για εθνικές συστάσεις πριν από την υποβολή στην κυβέρνηση και να προκαλεί συζήτηση και με την ε, κυβέρνηση της χώρας αυτής και με την αντιπολίτευση και ούτω καθεξής. Και να το κάνει αυτό και σε διάλογο και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πέραν αυτού, θεωρώ ότι οι εθνικές βουλές πρέπει να έχουν και ένα δικαίωμα υποβολής ερωτήσεων, περιορισμένο μεν, αλλά προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και ως αντάλλαγμα θεωρώ ότι θα πρέπει να δίνονται συγκεκριμένα στοιχεία στο, για το κάθε ευρωπαϊκό, ε, ευρωπαϊκό εξάμεινο που να είναι δεσμευτικά για την επίτευξη των στόχων της Ευρώπης 2020. Και όχι μόνο η Ευρώπη 2020, αλλά για κάθε ημερολογιακό έτος να προβλέπονται συγκεκριμένα δηλαδή ε, μέτρα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και για τις συγκεκριμένες σας προτάσεις. Ο Ιβο Ολιβέηρα έχει το λόγο από το Πορτογαλικό Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχει μεγάλη σημασία αυτή η συζήτηση μεταξύ κοινοβουλίων, γιατί ζούμε ε, μεγάλες αλλαγές έχει μεγάλη σημασία να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε την απασχόληση, πώς να αντιμετωπίσουμε τον αποπληθωρισμό και την κατανομή πλούτου. Έχει μεγάλη σημασία το πρόγραμμα επενδύσεων Juncker καθώς και ο πολλαπλασιαστικός παράγοντας. Όμως σε πολλές χώρες η κοινή γνώμη ζητά διαφορετική προσέγγιση, ιδιαίτερα όταν μιλάμε για τη ζωή των πολιτών. Βλέπουμε στην Πορτογαλία μεγάλη ανεργία των νέων, όπου ο παράγοντας της φτώχειας είναι πολύ υψηλός και ο τομέας της υγείας έχει καταβαραθρωθεί. Στα πλαίσια της λιτότητας υπάρχουν πολύ αρνητικές κοινωνικές επιπτώσεις. Οι νέοι έχουν μείνει πίσω. Η Επιτροπή μίλησε για μία νέα πρόταση υπέρ των νέων. Πρόκειται για έναν τομέα όπου υπάρχει κατεπίγουσα ανάγκη δράσης. Στην Ευρώπη 2020 μπορούμε να δράσουμε ταχύτερα μπορούμε να προβούμε σε μία επανακατανομή του πλούτου, έτσι ώστε οι νέοι να μπορέσουν να συμμετέχουν στο κοινωνικό γίγνεσθε και η Ευρώπη να γίνει πιο φιλική. Ευχαριστώ. Ο Στραν Τζούρκοβιτς έχει το λόγο από το Κοινοβούλιο της Κροατίας, αν προφέρα καλά το όνομά σας. Ναι, πολύ, πολύ καλά το ε, προφέρατε, Πρόεδρε. Και σας ευχαριστώ πολύ. Όταν μιλάμε για στρατηγικές και για την Ευρώπη 2020, το ζήτημα αυτό θα τύχει αναθεώρηση στα επόμενα χρόνια γιατί θα πρέπει να είναι ένας αποδοτικός μηχανισμός. Θα πρέπει να αναθεωρείται η κάθε μας στρατηγική γιατί υπάρχουν νέες προοπτικές και τάσεις. Μιλώντας για το ευρωπαϊκό εξάμεινο, θεωρώ ότι η δημοσιονομική εξυγίανση και η φορολογική σταθερότητα έχουν μεγάλη σημασία και οποιασδήποτε ανισότητες θα πρέπει να εξαλειφθούν. Αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι οι επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα και οι κυβερνήσεις θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα δραστήριες. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τη ρευστότητα των τραπεζών και τα χαμηλά επιτόκια που ισχύουν αυτή τη στιγμή. Όμως η αναμενόμενη ανάκαμψη δεν έλαβε χώρα και γι' αυτό ακριβώς ε, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο, να είναι δηλαδή κινητήριος δύναμη, να αποτελέσουν το κατάλληλο μηχανισμό μόχλευσης για να φτάσουμε σε συγκεκριμένες συνέργειες. Επίσης θα πρέπει να αναλύσουμε τη δυναμική του μηχανισμού συνεργειών για να δούμε πώς θα μπορέσουν να συνδράμουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή, γιατί έτσι μόνο θα φτάσουμε σε καλά αποτελέσματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο επόμενος, ο μιλτής ε, ε, Ρισάρ Γιούγκ από τη Γαλλική Γερουσία. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου πρώτα απ' όλα να εκφράσω την ικανοποίησή μου, μια που έχουμε ένα ποσοστό ανάπτυξης χαμηλό, υψηλή ανεργία και είμαστε μακριά για να μην μπω στα όρια του αποπληθωρισμού. Οπότε δύσκολο να είμαι και ενθουσιασμένος για όλα αυτά. Η συγκυρία είναι καλή, τα επιτόκια είναι χαμηλά, η τιμή του πετρελαίου είναι χαμηλή, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προχωράει σε μια πολιτική που ανταποκρίνεται στις επιθυμίες μας, συνεπώς πρέπει να πετύχουμε. Ένα από τα στοιχεία που αναφέρονται εδώ είναι το επενδυτικό πακέτο των 315 δισεκατομμυρίων. Αν η μόχλευση λειτουργήσει όπως είπαμε, είναι σαν τα 500 δις που θέλει να βάλει στις υποδομές η Αμερικανική κυβέρνηση. Πάντως, σίγουρα πρέπει να κάνουμε πιο γρήγορα. Το πρόβλημα δεν είναι το καθόμαστε και να συζητάμε για μήνες, για τη διακυβέρνηση, για τη μέθοδο. Το πραγματικό πρόβλημα είναι να επιλέξουμε σχέδια και να προχωρήσουμε. Γιατί οι επενδύσεις στο κάτω-κάτω αργούν να δώσουν αποτελέσματα στην πραγματική οικονομία. Ένα άλλο στοιχείο είναι ότι το επενδυτικό αυτό πακέτο πρέπει να χρησιμεύσει σε κοινέ πολιτικέ, σε πολιτικέ δηλαδή που να εξυπηρετούν την ολοκλήρωση τη ενία αγορά και την ολοκλήρωση τη Ευρώπη. Τα δίκτυα, ενέργεια κλπ. κλπ. Ζητώ λοιπόν και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από τις χώρες μέλη να πάμε πιο γρήγορα για τις, στις αποφάσεις και στην εφαρμογή τους όσον αφορά αυτό το επενδυτικό πακέτο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ιβάνα Μαλέτιτς από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τώρα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Καλησπέρα σε όλους σας. Θέλω να υποδεχτώ εδώ τους συναδέλφους από τα Εθνικά Κοινοβούλια και τους άλλους ευρωβουλευτές. Είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε πόσο κοντά και πόσο μακριά συγχρόνως βρισκόμαστε από τους στόχους της στρατηγικής 2020 σε σχέση με τη στιγμή που αποφασίστηκαν οι στόχοι αυτοί. Ενισχύσαμε την απασχόληση, μειώσαμε την ένδια, αυξήσαμε τον αριθμό του πληθυσμού που έχει μεγάλη μόρφωση. Προχωρήσαμε όσον αφορά την αυτονομία μας από τους ενεργειακούς πόρους, όσον αφορά το ποσοστό του ΑΕΠ που επενδύουμε στην ανάπτυξη. Αυτά είναι τα ερωτήματα που πρέπει να υποβάλουμε σε αυτούς μας. Και ένα άλλο είναι το κατά πόσο η στρατηγική στις επιμέρους χώρες έδωσε κάποια αποτελέσματα σε σχέση με τους στόχους του 2020. Η στρατηγική αυτή 2020 ετοιμάστηκε τελικά βάσει στόχων που να έχουν να κάνουν πράγματι με την εθνική στρατηγική. Πώς θα πετύχουμε τους στόχους. Το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο πρέπει να χρησιμοποιήσει τις συστάσεις προς τις χώρες για να συντονίσουν τις δραστηριότητές τους προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι των στρατηγικών κειμένων. Χρειάζεται υψηλό επίπεδο σύνδεσης με τα έγγραφα αυτά. Επιπλέον, η συνοχή, η γεωργική πολιτική είναι υπεύθυνε για ένα μεγάλο μέρος του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού και χρειάζεται βέβαια καλό συντονισμό στα πλαίσια του ευρωπαϊκού εξαμήνου, αλλιώς δεν θα πετύχουμε τους στόχους μας για επένδυση και οικονομική ανάπτυξη. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Επόμενος ομιλητής. Ανδρέας Καλασεύσκη. Από το Κοινοβούλιο της Πολωνίας, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρόεδρε, εδώ και μερικά χρόνια Ζήσαμε μια μεγάλη αποτυχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα θα πρέπει να υλοποιηθεί η στρατηγική της Ευρώπης 2020. Ένα πολύ βασικό έγγραφο και έχει μεγάλη σημασία να κριθεί ως ευέλικτο μέσο. Αν δεν είναι ευέλικτο, τότε θα αντιταχθεί στην πραγματική ανάπτυξη, την οποία επιθυμούμε. Γι' αυτό πριν υποχρεώσουμε ορισμένα κράτη-μέλη να δράσουν, θα ήταν καλύτερα να δούμε κατά πόσο αυτό το έντυπο είναι ε, πραγματικά ένα σκόπιμο εγγραφό, κατά πόσο δηλαδή δεν πρέπει να γίνει μία αναθεώρηση από τους πολιτικούς, για να μην είμαστε ιδιαίτερα άτεγκτοι και να μην περιοριστούμε σε δόγματα. Έχουμε πολλές πολιτικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο, συνοχής, δημοσιονομική, φορολογική. Αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε κατά πόσο οδηγούν σε μια πραγματική ανάπτυξη. Υπάρχει και ένα άλλο σημαντικό στοιχείο. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει έναν προϋπολογισμό με συνεισφορά που υπερβαίνει κατά τι το 1% από το εθνικό ΑΕΠ. Άρα το 90% βρίσκεται στα χέρια των εθνικών προϋπολογισμών. Άρα είμαστε πολύ περιορισμένοι ως προς το περιθώριο ελιγμών. Γι' αυτό θα πρέπει οι επιδοτήσεις και οι πιστώσεις να δαπανώνται σωστά για να υπάρχει πραγματικά προστέμενη αξία για κάθε ευρώ που ε, δαπανάτε. Αυτό επίσης που έχει εντύπωση είναι να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε και την απασχόληση με νέες θέσεις εργασίας και με τα έσοδά μας. Δεν πρέπει να ξεχνάμε τη δυναμική του ιδιωτικού τομέα και τη συμμετοχή του. Η διοίκηση είναι πολύ δημιουργική στη δημιουργία προσκομμάτων και εμποδίων περισσότερο από κάθε άλλο. Ας αφήσουμε να αναπνεύσει ο επιχειρηματικός κόσμος για να προχωρήσουμε πραγματικά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο Παύλος Σά από την Πορτογαλία. Ευχαριστώ πρόεδρε, κύριε πρόεδρε, κύριοι βουλευτές του Ευρωκοινοβουλίου και των Εθνικών Κοινοβουλίων. Μιλήσαμε για τους στόχους της στρατηγικής Ευρώπη 2020 για να έχουμε καλή και ποιοτική εργασία. Όμως ε, υπάρχουν πολλές αντιφάσεις με το πρόγραμμα της Τρόικας που εφαρμόστηκε στην Πορτογαλία τα τελευταία τρία χρόνια. Τι συνέβη σε σχέση με την αγορά εργασίας. Είδαμε ότι έχασαν την εργασία τους χιλιάδες άνθρωποι. Ανήλθε η ανεργία σε ιστορικά υψηλά όρια, ιδιαίτερα μεταξύ των νέων δεν είχαμε συλλογικές συμβάσεις, είχαμε κακοπληρωμένες εργασίες και μετανάστευση των νέων που δεν έβρισκαν καμία προπτική εργασία στην Πορτογαλία. Ε, μας σοκάρει το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ανακοίνωση 902 του Δεκεμβρίου 2014 μίλησε για υποδειγματικές μεταρρυθμίσεις στην Πορτογαλία. Η στρατηγική της Λισαβόνας εγκρίθηκε εδώ και 15 χρόνια και τότε οι πολιτικοί ηγέτες μίλησαν για διασφάλιση της εργασίας. Ε, ελέγχθη τότε ότι το 2010 θα, η Ευρώπη θα είναι η πιο ανταγωνιστική ήπειρο στον κόσμο με έλλειψη οποιασδήποτε μορφής κοινωνικού αποκλεισμού. Δυστυχώς όμως η φτώχεια άγγιξε το 20% του πληθυσμού και ένα από κάθε τρία παιδιά ζουν σε μια φτωχή οικογένεια. Άρα η στρατηγική 2020 δεν βοήθησαν τους εργαζόμενους, αλλά τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα. Έτσι είχαμε μια επιδίνωση της εκμετάλλευσης θα πρέπει να έρθουμε σε ρήξη με αυτές τις πολιτικές και να επιβάλλουμε πολιτικές που έχουν προτεραιότητα την απασχόληση και την κοινωνική συνοχή έτσι ώστε να εγγυηθούμε τα δικαιώματα των εργαζομένων. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Τώρα δίνω το λόγο στον Σωτήρη Τζαριανόπουλο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και δίνω το αναθέτω Προεδρία στην Μαρίτα Ουλσβοκ, Αντιπρόεδρο τη Επιτροπής Απασχόλησης. Στις εκλογές άναψε κυριολεκτικά η συζήτηση για τις υπερχρεωμένες χώρες. Γαλλία, Ιταλία, Ελλάδα και η νευαρχίδα του υπεριαλισμού Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής που ξαφνικά δίθεν αγάπησαν τον ελληνικό λαό ανταγωνίζονται για τη Γερμανία, όχι για τα λαϊκά συμφέροντα, αλλά για τους όρου πληρωμής ενός χρέους που δεν χρωστάνε οι λαοί. Ανάπτυξη εννοείται η ελεημοσύνη στην ακραία φτώχεια και δισεκατομμύρια από την άλλη στα μονοπόλια με ποσοτική χαλάρωση του Ντράκη με επενδυτικά πακέτα του Γιούγκερ. Μπορεί η Τρόικα και τα μνημόνια να αλλάξουν όνομα, όχι όμω ουσία. Όλε οι πλευρέ παρά του ανταγωνισμού του συμφωνάνε στη λέξη κλειδί. Διαρθρωτικέ μεταρρυθμίσει, Δηλαδή, μείωση φόρων για τι επιχειρήσει και άλλη μείωση, περισσότεροι ακόμα φόροι για το λαό Μόνο έτσι μπορούν να προκύψουν οι σοσκελισμένοι προπολογισμοί που είναι ο στόχο τη πολιτική αυτή. Και από την άλλη, μείωση του εργατικού κόστου, γενίκευση τη ευέλικτη εργασία, περαιτέρω χτύπημα τη κοινωνική ασφάλιση για την ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων. Αυτά λέει το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και η στρατηγική του 2020. Δηλαδή τα μνημόνια διαρκείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι εδώ με βάση αυτά διαπραγματεύεται και η νέα ελληνική κυβέρνηση που τα σέβεται και τα στηρίζει θερμά. Οι λαοί όμως δεν μάτωσαν για ψίχουλα. Η ανάκτηση των απολειών τους σημαίνει σύγκρουση και αποδέσμευση με την, Ευρωπαϊκή Ένωση, μονομερή διαγραφή του χρέους και κοινωνικοποίηση των μονοπωλίων. Thank you. Κυρία ευχαριστώ. Πάολο Γκερέρι, Ιταλός. Ας αναγνωρίσουμε ότι δεν έχουν επιτευθεί στόχοι ως τώρα της στρατηγικής 2020, βέβαια για διάφορους λόγους, αλλά πρέπει να αναγνωρίσουμε όμως και ορισμένα θεμελιώδη σφάλματα στην διατύπωση και στην εφαρμογή της στρατηγικής αυτής. Έχουν γίνει τα σφάλματα αυτά. Νομίζω λοιπόν ότι η διάμεση αυτή επανεξέταση θα πρέπει να δώσει την ευκαιρία μιας ριζοσπαστικής αναθεώρησης στρατηγικής και ιδίως πώς να διασυνδεθεί η στρατηγική 2020 με το ευρωπαϊκό εξάμεινο που μέχρι τώρα αυτά τα πράγματα ήταν χωρισμένα. Από αυτή την άποψη υπάρχει και η ευκαιρία να ενισχυθούν οι στόχοι του εξαμήνου, ιδίως αν επιθυμούμε να προωθήσουμε στα σοβαρά μια στρατηγική ανάπτυξης βασισμένη σε επενδύσει πάνω σε τρεις άξονες. Πρώτα, το περιεχόμενο της Ευρώπης 2020 είναι σαφές ότι η στοχοθέτηση στο ευρωπαϊκό επίπεδο και η μεταφορά των στόχων σε δράσεις που θα υιοθετηθούν στο εθνικό επίπεδο, αυτό λοιπόν δεν έχει λειτουργήσει αυτό που θα μπορούσαμε να κάνουμε λοιπόν τώρα θα ήταν να βάλουμε κάποιους στόχους για μεγαλύτερη οικονομική ολοκλήρωση στο ευρωπαϊκό επίπεδο, έτσι ώστε να έχουμε πανευρωπαϊκούς στόχους, που θα είναι κάτι παραπάνω από ένα άθροισμα των εθνικών στόχων. Από την άποψη αυτή είναι καθαρό ότι, για παράδειγμα, στον χώρο των υποδομών ενό είδου δηλαδή πανευρωπαϊκών υποδομών. Είναι ένα πολύ σημαντικό στόχο που μπορεί να μπει στο επίκεντρο τη νέα αυτή προσπάθεια. Δεύτερο, η διαχείριση αυτή τη στρατηγική. Αυτό ήταν πάντα το αδύναμο σημείο της Ευρώπης 2020 για διάφορους λόγους όπως η εξέταση από τους ομοτήμους, η αμοιβαία δηλαδή, ο έλεγχο και ούτω δεν επέτυχε, διότι υπήρχε μια μεγάλη απόσταση ανάμεσα σε αυτή την προσέγγιση και στην προσέγγιση του εξαμήνου και τη σταθερότητα του εξαμήνου κτλ. Από αυτή την άποψη λοιπόν η προσπάθεια να διασυνδεθούν τα δύο βρίσκω ότι είναι πολύ σημαντικό για παράδειγμα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ετήσια επισκόπηση ανάπτυξης να αναφερθεί ειδικά στην πρόοδο που είναι αναγκαία για την επίτευξη των στόχων της ε, Ευρώπης 2020, που τώρα δεν έχει γίνει. Τρίτο, αν μπορέσουμε να αλλάξουμε το περιεχόμενο και να αναθεωρήσουμε τη διαχείριση, governance δηλαδή, θα είναι δυνατό νομίζω να επανατοποθετήσουμε τη στρατηγική μέσα στα πλαίσια μιας ευρωπαϊκής στρατηγικής. Από την άποψη αυτή είναι καθαρό ότι Υπάρχει αυτή η διάκριση ανάμεσα σε αυτά που μπορούμε να ορίσουμε σαν καθορισμό, σαν πρόταση μάλλον νέων κανόνων στο ευρωπαϊκό επίπεδο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με, τον με τους μακροπρόθεσμους στόχους. Είναι δύο διαφορετικά επίπεδα, πάρα πολύ όμως διακεκριμένα μέχρι τώρα, με μεγάλη απόσταση μεταξύ τους. Πρέπει να δούμε ποια διασύνδεση μπορούμε να αποκαταστήσουμε εδώ. Από αυτή την άποψη δηλαδή με αναθεώρηση και το περιεχόμενο αναθεώρηση και της διαχείρισης μπορούμε να επανατοποθετήσουμε τη στρατηγική στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής προσπάθειας δίνοντας έτσι τη δυνατότητα να ενισχύσουμε τις δράσεις και πάλι για να ξεκινήσει η ανάπτυξη στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Ευχαριστώ κύριε Ολσκόλ. Η κυρία Καβριέλα Κρέτσου από τη Ρωμανία. Αγαπητοί συνάδελφοι, η στόχοι είναι πολύ καλή. Το πώς θα τους επιτύχουμε είναι κάτι το διαφορετικό. Στη Ρώμη την ε, πρώτη μέρα μιλήσαμε κατά τη διάσκεψη αυτή για την επικινδυνότητα του δημόσιου χρέους και πώς θα πρέπει να αποφύγουν οι κυβερνήσεις να συνάψουν νέα χρέη. Τη δεύτερη ημέρα μιλήσαμε για το πιστοτικό πλαίσιο και την εμπιστοσύνη του χρηματοοικονομικού τομέα. Υπάρχει καλό και κακό χρέος δηλαδή. Άρα ανέκυψε μια νέα ιδέα. Υπάρχουν κακές επενδύσεις που προέρχονται από το δημόσιο άμεσα και που στην ουσία υποσκάπτουν την ε, δημοσιονομική εξυγίανση και οι καλές επενδύσεις αυτές του ιδιωτικού τομέα. Έτσι αναφέρθηκε, μα αυτό είναι ιδεολογικό ζήτημα. Δεν αφορά με την ε, οικονομική πολιτική. Η, η ιδεολογία δεν είναι κακή αυτή καθεαυτή, αλλά βλέπουμε ότι δεν φτάσαμε σε αυτά αποτελέσματα. Ήταν πολύ αδύναμα τα αποτελέσματα. Γιατί αρνείστε τις δημόσιες άμεσες επενδύσεις και την αύξηση της ζήτησης και την καταπολέμηση των ανισοτήτων για να ανορθώσουμε την οικονομία. Γιατί το αρνούνται αυτό οι Ευρωπαίοι πολιτικοί. Μία μεγαλύτερη ζήτηση θα ανόρθωνε την εμπιστοσύνη του κοινού. Δυστυχώς όμως δεν το καταφέραμε. Θα πρέπει άμεσα να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα και ως δημοκρατικό όργανο. Ο κύριος Πυρίνσκι από τη Βουλγαρία, Ευρωβουλευτής, έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, στην δήλωση της Επιτροπής Μπαρόσο πριν από ένα χρόνο περίπου, το Μάρτιο δηλαδή που μας πέρασε, αναφέρεται σαφώς ότι κατά το παρελθόν η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν ένας μηχανισμός που μείωνε τις διαφορές. Τώρα όμως με την κρίση οι διαφορές μεγαλώνουν και μεταξύ χωρών αλλά και μέσα στις ίδιες χώρες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο ίδιο κείμενο λέει ότι θα υπάρξει δημόσια κρόαση και ότι θα γινόταν στα τέλη της προηγούμενης χρονιάς, ώστε στις αρχές του 2015 να μπορούμε να έχουμε τη μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση για να αλλάξουμε και τους στόχους και τις πολιτικές ενδεχόμενα. Εξεπλάγει λίγο από αυτά που άκουσα από τον κύριο Κατάινεν, γιατί είπε ότι υπάρχουν πολλά άλλα που πρέπει να γίνουν και γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναβάλλει τη μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση. Ναι, αλλά η νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή Πώς θα σχεδιάσει το επενδυτικό ταμείο χωρίς προηγουμένως να γνωρίζει το τι έχει γίνει μέχρι τώρα στην εφαρμογή της στρατηγικής της και τι αλλαγές χρειάζονται. Επίσης πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχασε μια ευκαιρία. Έχασε την ευκαιρία να συνδέσει την αναθεώρηση αυτή σε επίπεδο Ευρώπης, Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και συγχρόνως να υπάρχει αναθεώρηση και από τα Εθνικά Κοινοβούλια στα εθνικά προγράμματα βάσει της στρατηγικής. Τότε θα μπορούσαμε συντονισμένα να έχουμε στόχους και περισσότερα κίνητρα για τη δεύτερη φάση εφαρμογής της στρατηγικής μας. Το πρόβλημα που αναφέρει η Επιτροπή στην έκθεσή της είναι σοβαρό, γιατί αρχίζουν από τις κοινωνικές συνέπειες της κρίσης, που είναι επίσης το θέμα της γύρανσης του πληθυσμού, το κατεξοχήν πρόβλημα που έχει πάρα πολλές συνέπειες στην απασχόληση, στις κοινωνικές πτυχές κτλ. Και ένα άλλο κοινωνικό ζήτημα είναι οι αυξανόμενες κοινωνικές ανισότητες. Υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα σε αυτούς που έχουν τα υψηλότερα εισοδήματα και αυτούς που έχουν τα χαμηλότερα. Το χάσμα μεγαλώνει. Θα ολοκληρώσω δηλώνοντας την πεποίθησή μου, τη βαθιά μου πεποίθηση, που είναι ότι η Επιτροπή Juncker δεν ξέρει ακριβώς τι πρέπει να κάνει, δεν έχει τη βούληση ούτε την επιθυμία να λύσει τα προβλήματα προσπαθεί απλώς βραχυπρόθεσμες λύσεις να, βρεις, να βρει για να δείξει ότι κάτι κάνει. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, ευχαριστούμε κύριε Πυρίνσκι. Το λόγο έχει τώρα η Περβάνς Μπερές, Ευρωβουλευτής. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητή Πρόεδρε. Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, ο Αλεξάνδερ Σάμπα αναφέρθηκε στα δικηδεύματα της εσωτερικής αγοράς. Εγώ θέλω να επανέλθω σε κάποιες πτυχές που δεν αναφέρθηκαν για το σχέδιο Juncker. Μιλάμε πάντα για την εσωτερική αγορά όταν μιλάμε για το επενδυτικό πακέτο Juncker. Αν όμως θέλουμε οι μακροχρόνιες επενδύσεις να χρηματοδοτήσουν και τις οικολογικές αλλαγές που αποτελούν ένα σημαντικό άξονα του σχεδίου Juncker, τότε η τιμή του άνθρακα είναι ζωτική σημασία. Δεν θα υπάρχουν μακροχρόνιε επενδύσεις στην προστασία του περιβάλλοντος αν δεν φροντίσουμε για την τιμή του άνθρακα. Ακόμα δεν υπάρχει συμφωνία για να τεθούν σε εφαρμογή αποφάσεις μας προκειμένου να σταθεροποιηθεί και να είναι προβλέψιμη η τιμή του άνθρακα. Αυτό ήταν το πρώτο. Δεύτερον, για την ψηφιακή διάσταση του επενδυτικού πακέτου Juncker. Υπάρχει πτυχή εσωτερική αγορά ζωτική σημασία και αυτή. Και ελπίζω με τα εθνικά κοινοβούλια να μπορέσουμε να κινητοποιηθούμε. Διότι σε τι θα μας βοηθούσε να έχουμε μαζική επένδυση υπέρ της ψηφιακής οικονομίας αν οι επιπτώσεις των επενδύσεων αυτών δεν κατέληγαν στους κύριους ε, δικαιούχους, στους ε, φυσιολογικούς δικαιούχους που πιάλι είναι οι Ευρωπαίοι πολίτες. Αν Δηλαδή καταλήξουν τα κέρδη στη Facebook και στην Amazon. Χρειάζονται λοιπόν ναι, επενδύσεις στη ψηφιακή αγορά, αλλά συγχρόνως πρέπει να επενδύσουμε και στην φορολογία αυτού του είδους της νέας οικονομίας που ξεφεύγει από τη φορολογία προς το παρόν. Και τρίτον, θέλω να ευχαριστήσω πολύ τους συναδέρφους, μάλλον τον συνάδελφο, τον κύριο Σαραζάν από την Bundestag, που στήριξε προτάσεις που και εμείς πιστεύουμε ότι είναι πολύ σημαντικές για να διατηρηθεί ζωντανή δημοκρατία στην Ευρώπη. Την συναπόφαση όσον αφορά την ετήσια επισκόπηση για την ανάπτυξη και τις συστάσεις αναχώρα. Νομίζω ότι εδώ η συνεργασία μας μπορεί να είναι ιδιαίτερα καρποφόρος. Ευχαριστούμε κύριε Πέρες. Το λόγο έχει τώρα ο κύριος Νοφίτου. Κύπρος. Thank Συζητάμε τους τρόπους για να βγούμε από την ύφεση και όλοι συμφωνούμε πως ο δρόμος είναι μέσα από την ανάπτυξη. Είναι σημαντικό το πακέτο του Πρόεδρου Γιούγκερ των 315 δισεκατομμυρίων όπως και πολύ σημαντική η απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για την ποσοτική χαλάρωση. Αλλά φοβούμε ότι αυτά από μόνα τους δεν είναι αρκετά. Την οικονομική ανάπτυξη σε μια ελεύθερη οικονομία όπως είναι και η ευρωπαϊκή μπορούμε να την πετύχουμε μέσα και μόνο από ιδιωτικές επενδύσεις. Και ξεχνάμε και είναι εκτός της συζήτησής μας το κυριότερο κατά την άποψή μου πρόβλημα που έχουμε στην Ευρώπη εδώ και χρόνια η ευρωπαϊκή οικονομία έχει απολέσει την ανταγωνιστικότητά της. Δεν είναι πλέον ανταγωνιστική. Γι' αυτό και δεν υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για επενδύσεις. Και πρέπει για να μπορέσουμε να ξανακερδίσουμε την ανταγωνιστικότητα πρέπει να λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στην Ευρώπη Έχουμε μια Ευρώπη υπερχρεωμένη, μια γυράσκουσα Ευρώπη με γυρασμένο πληθυσμό, μια Ευρώπη που έχει έλλειψη ενεργειακών πόρων αλλά συνάμα αντιμετωπίζει και το θέμα της ενεργειακής ασφάλειας μια Ευρώπη που είδε αρκετές από τις βιομηχανίες της να ξενιτεύονται σε τρίτες χώρες και την ίδια ώρα χάσαμε εδώ και καιρό τη μάχη της ψυχτιακής οικονομίας. Άρα αν δεν διορθώσουμε αυτά τα προβλήματα, αν δεν αποκτήσουμε την ανταγωνιστικότητα στην ευρωπαϊκή οικονομία, θα μιλούμε για αρκετά ακόμα χρόνια για τα προβλήματα της ύφεση. Και θέλω να το διευκρινίσω, προέρχομαι από μια χώρα που έχει δεχτεί ένα σκληρό μνημόνιο, δεν είμαι όμως εξ εκείνων που πιστεύω πως μπορούμε να κερδίσουμε την οικονομική ανάπτυξη με περισσότερα δανεικά. Δεν μπορεί να είναι βιώσιμη η οποιαδήποτε ανάπτυξη με το να συνεχίζεις να δανείζεσαι. Πρέπει να κάνουμε την ευρωπαϊκή οικονομία ανταγωνιστική και να νοικοκυρεύσουμε τα δημόσια οικονομικά. Thank Πρόεδρος ευχαριστώ. Η Ευρωβουλευτής από την Πορτογαλία. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ένα από τα ζητήματα που μας απασχολεί όταν μιλάμε για δημιουργία νέων θέσεων εργασίας είναι το πώς ζουν οι εργαζόμενοι σήμερα. Στη χώρα μου και όχι μόνο στην Πορτογαλία αναφέρεται ότι κάθε φορά είναι υψηλότερος ο αριθμός των εργαζομένων, αλλά αυξάνεται συνάμα και η φτώχεια. Όταν μιλάμε λοιπόν για επενδύσεις, θα πρέπει να ρωτήσουμε σε ποιους απευθύνεται, ποιους αφορά βεβαίως τονώνει την οικονομία, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι η ευημερία των ανθρώπων. Έτσι μόνο έχει νόημα ένα επενδυτικό πρόγραμμα. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι δεν υπάρχει καμία ρήτρα διασφάλισης σε αυτό το σχέδιο σε σχέση με σταθερή απασχόληση και όχι επισφαλή. Μιλάμε για υποδομές, ιδιαίτερα στον τομέα της ενέργειας και των μεταφορών, όπου οι μόνοι κερδισμένοι είναι οι μεγάλες κοινοπραξίες. Όμως, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι οι θέσεις εργασίας, ασφαλούς εργασίας, μη επισφαλούς, αξιοπρεπούς εργασίας, ιδιαίτερα για αυτούς που βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας. Θα ήθελα να υποβάλω δύο ερωτήματα σε σχέση με την ετήσια έκθεση της Επιτροπής για το 2015. Πρόκειται για δύο προτάσεις. Όταν λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι μας ενδιαφέρει το επίπεδο των κοινωνικών παροχών και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη δημιουργία θέσεων εργασίας και προβολής κοινωνικών παροχών. Θα ήθελα να ρωτήσω τι εννοείτε. περισσότερα στάζ, σταθερή εργασία, συμβασιούχους. Στην ουσία, αν πρόκειται για κάτι τέτοιο, δεν επιλύεται το θέμα της απασχόλησης, διότι αν γίνει αυτό που γίνεται μέχρι σήμερα, όπου απολύονται χιλιάδες δημόσιοι υπάλληλοι στη χώρα μου και παράλληλα ε, προκυρήσονται συμβάσεις ορισμένου χρόνου και στάς, τι κάνουμε. Δεν κάνουμε τίποτα άλλο από το να αυξάνουμε την επισφάλεια, διότι πρόκειται για θέσεις εργασίας που δεν είναι μόνιμες. Άρα αυτό που έχει σημασία είναι τα κοινωνικά κονδύλια να χρησιμεύσουν πραγματικά για θέσεις εργασίας, όχι θέσεις επισφαλούς εργασίας. Επίσης, θα ήθελα να πω ότι δεν μπορεί η Κομισιόν να παρεμβαίνει στις συλλογικέ συμβάσεις και στο εργατικό δίκαιο των κρατών μελών. Δηλαδή δεν μας ενδιαφέρει να υπηρετούμε την εργοδοσία. Γιατί η Επιτροπή παρεμβαίνει σε εθνικά ζητήματα και ιδιαίτερα στις συλλογικές συμβάσεις, γιατί δεν προωθεί την πραγματική ισότητα μεταξύ ανθρώπων και γυναικών. Νομίζω ότι έχει σημασία να δούμε ποια είναι τα συμφέροντα που υπερασπίζεται η Επιτροπή όταν προβάλλει συγκεκριμένες θέσεις. Ο κύριος Αρτουή έχει το λόγο, ο πρόεδρος της Επιτροπής Προϋπολογισμών. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Προσοχή στις χήμερες. Η στρατηγική της Λισαβόνας, για παράδειγμα, ήταν πάρα πολύ ωραία. Και έτσι με μια καλή χειρονομία, οι ηγέτες κατό και κυβερνήσεων ενέκριναν τη στρατηγική αυτή είναι όμως η αντίθεση ανάμεσα στους στόχους της και τις πράξεις που έκαναν οι περισσότερες κυβερνήσεις δηλαδή. Το ίδιο μπορούμε να πούμε τώρα για τη στρατηγική του 2020. Έχουν ανακοινωθεί πολύ ωραία πράγματα. Εξάλλου ο κύριος Κατάινεν είπε ότι θα δημιουργήσουμε πολλές θέσεις απασχόλησης με το επενδυτικό πακέτο Juncker. Αλλά εγώ θυμάμαι αυτά τα οποία δηλώναμε όταν άρχισε να κυκλοφορεί το ευρώ. Είπαμε ότι η Ευρωζώνη θα γίνει η πιο ευημερούσα περιοχή του κόσμου. Και πού βρισκόμαστε σήμερα. Το πρόβλημα κατά τη γνώμη μου είναι η διακυβέρνηση στην Ευρώπη ή πιο σωστά η απουσία κυβέρνησης με όλα τα αποτελέσματα που έχει αυτό. Η Ευρωζώνη δεν ήταν παρά το πρώτο θύμα λειτουργήσε αρκετά καλά για 10 περίπου χρόνια. Το είπαμε αυτό στον απολογισμό μας. Δύο παρατηρήσεις όμως έχω να κάνω τώρα. Σήμερα το πρωί συνεδρίασε η Επιτροπή μας με θέμα τις οφειλές, τους απλήρωτους λογαριασμούς. Η Ευρώπη δημιουργεί οφειλές γιατί δεν τιμά τις υποχρεώσεις της, δεν πληρώνει τους λογαριασμούς για τους οποίους έχει αναλάβει τη δέσμευση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν πληρώνει γιατί δεν διαθέτει τα μέσα και έτσι συσσωρεύεται η οφειλή. Τι πρέπει να κάνουμε αμέσως, πώς θα ευαισθητοποιήσουμε τις κυβερνήσεις. Το φθινόπωρο του 2014 επίσης το συζητήσαμε. Και υπήρχε ένας απρόβλεπτος πόρος μάνα εξ ουρανού και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπόρεσε να εισπράξει 5 δισεκατομμύρια από πρόστιμο. Εμείς είχαμε σκεφτεί ότι τα 5 αυτά δισεκατομμύρια θα έπρεπε κατά προτεραιότητα να πάνε στην πληρωμή των πιο παλιών λογαριασμών που χρωστάγαμε. Οι κυβερνήσεις όμως αποφάσισαν να πάρουν τα 5-7 δισεκατομμύρια πίσω για να βελτιώσουν, είπανε, την κατάσταση στους προπολογισμού τους. Τελικά όμως οι απλήρωτοι αυτοί λογαριασμοί είναι οφειλέ των χωρών μελών. Και αν ήταν εδώ ακόμα ο κύριο Κατάινεν θα του πρότεινα όταν θα εξετάσει τους ετήσιους λογαριασμούς των χωρών μελών να προσθέσει στη, στα χρέη των χωρών μελών και το κομμάτι εκείνο που τους αναλογεί από τις οφειλές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορεί να ακούγεται προκλητικό αυτό, αλλά πρέπει να είμαστε πιστοί στην εικόνα τελικά των ε, λογαριασμών μας. Έπειτα για τη στρατηγική 2020, Η πρόεδρος της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων ε, του Πολωνικού Κοινοβουλίου μας είπε ότι το χρέος μας είναι 1% του ΕΠ. και ότι οι οικονομίες είναι των χωρών μελών. Ότι δεν χρειάζεται να σκεφτούμε εναρμόνιση είπε στους λογαριασμούς που κάνουν οι χώρες μέλη για την ε, αξιολόγηση της ειλικρίνειας των λογαριασμών, ότι αρκεί να προσθέσουμε τους λογαριασμούς αυτούς για να καταλήξουμε στο συμπέρασμα το τι είναι ο προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άρα και το χρέος της. Ο συντονισμός των Υπουργών χρειάζεται για να έχουμε περισσότερη ανάπτυξη και να αντιμετωπίσουμε καλύτερα την ανεργία. Θέλω να πω για τους ίδιους πόρους εδώ ότι είμαστε ανυπόμονοι. Περιμένουμε τις προτάσεις Μόντι, της ομάδας Μόντι δηλαδή. Αλλά φοβάμαι ότι δεν είναι ό,τι πιο εύκολο. Και δεν θα μπορέσουμε να καταλήξουμε χωρίς τη συνδρομή των Εθνικών Κοινοβουλίων. Υπάρχουν τόσες διαφορές στις διοικητικές συνήθειες, στην οτροπία. Ένας τέτοιος φόρος δεν θα απέδιδε το ίδιο σε όλες τις χώρες. Αλλά θα ήθελα να αρχίσουμε να το σκεφτόμαστε. Νωρίτερα αναφερθήκαμε στον άνθρακα, στη τιμή του άνθρακα. Ο φόρος στον άνθρακα που θα συλλέγαμε στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μήπως θα μπορούσε να χρηματοδοτήσει καλά τον προπολογισμό μας και θα μείωνε την εισφορά των χωρών μελών. Μήπως θα ήταν μια απάντηση αυτό για να πληρωθούν οι απλήρωτοι λογαριασμοί, οι οφειλές μας. Αν πάντως θέλουμε να πετύχει η οικονομική μας πολιτική, με την διακυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα γίνει αυτό, που τώρα τόσο πολύ λείπει. Δυστυχώς. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Κώστας Μαυρίδης τώρα, Κύπρος, Ευρωβουλευτής. Παρακαλώ. Θα ξεκινήσω με μια επισήμανση που αφορά στρατηγική, την Ευρωπαϊκή Στρατηγική 2020. Το περιεχόμενο της δεν, είναι, δεν αφορά μόνο ένα οικονομικό μοντέλο. Το περιεχόμενο της δεν αφορά μόνο ένα κοινωνικό μοντέλο. Αφορά και τα δύο Γι' αυτό όταν μιλάμε πρέπει να το έχουμε αυτό υπόψη μας. Είναι οικονομικό και ταυτοχρόνως υπάρχουν και κοινωνικές επιδιώξεις. Δύο διαπιστώσεις. Διαμορφώθηκε αρχικώς σε σαφώς διαφορετικές συνθήκες από τις σημερινές. Έχουν προκύψει φοβερές ανατροπές μέσα στην οικογένειά μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει λοιπόν να ληφθούν και αυτά υπόψη. Δεύτερον, οι στόχοι, όπως σωστά έχει λεχθεί από διάφορους συναδέλφους, δεν έχουν επιτευχθεί. Και θέτω ένα ερώτημα προς όλους μας. Είναι κάποιος εδώ που μπορεί με αυτοπεποίθηση να δηλώσει ότι οι στόχοι όσον αφορά και το κοινωνικό και το οικονομικό μοντέλο θα επιτευχθούν στα επόμενα χρόνια. Νομίζω θα συμφωνήσουμε ότι δεν το πιστεύουμε με αυτοπεποίθηση. Και ρωτώ λοιπόν, οι Ηνωμένε Πολιτείε που μπήκαν σε αυτή την κρίση πολύ πριν από εμάς, πώς βρίσκονται σήμερα σε σαφώς καλύτερη θέση από εμάς. Μπορούμε να μιλούμε για ώρες, αλλά πρέπει να παραδεχτούμε ότι τουλάχιστον ακολούθησαν μια εντελώς διαφορετική μακροοικονομική πολιτική. Εμείς προσπαθούμε ακόμα να την ακολουθήσουμε με το σταγονόμετρο και με πολύ χρονική υστέρηση. Και κάτι τελευταίο. Επενδυτικό πακέτο Juncker. Έχει γίνει παραδεχτό από τα δεξιά μέχρι τα αριστερά ότι χωρίς δημόσιο χρήμα δεν βγαίνουμε από αυτή την κρίση. Και πολύ σωστά. Τονίζω όμως και το εξής. Γιατί πρέπει να φτάσουμε στα όρια της, της απόγνωσης σε ορισμένα μέλη της οικογένειάς μας, της ευρωπαϊκής, για να προβούμε ή να μελετήσουμε έστω σημαντικές αλλαγές. Έπρεπε να φτάσουμε μέχρι εδώ για να σκεφτούμε ότι είναι καιρός να εγκαταλείψουμε την Τρόικα και να την υποκαταστήσουμε με δικά μας ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Σας ευχαριστώ. Ε, Η πρόεδρος Hayden από την Ιρλανδία. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να τοποθετηθώ. Η αναθεώρηση της στρατηγικής 2020 είναι επίκαιρη. Νομίζω ότι χρειάζεται να δοθεί λίγη περισσότερη προσοχή στις περιφέρειες. Υπάρχει άποψη ότι η σημερινή στρατηγική ακολουθεί μια προσέγγιση one size fits all. Δεν λαμβάνει υπόψη τις περιφερειακές διαφορές μεταξύ χωρών μελών. Όμως για να αποδοθούν οι αυξανόμενες ανισότητες πρέπει να ληφθεί υπόψη. Άκουσα τα σχόλια της Ρουμάνας συναδέλφου προηγουμένως σχετικά με το μέσο εισόδημα των Ρουμάνων σε σύγκριση με το συνολικό ευρωπαϊκό επίπεδο. Βεβαίως και υπάρχουν περιφερειακά θέματα, όμως δεν φαίνεται να λαμβάνονται παρκώς υπόψη. Σκέφτομαι ότι και η στατική 2020 θα εξακολουθήσει να μην πετυχαίνει τους στόχους εάν εξακολουθήσει να είναι μια διαδικασία από πάνω προς τα κάτω και όχι συμπεριληπτική. Πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στις συνεργασίες. Ιδίω για την φτώχεια δεν έχει πετύχει τίποτα στρατηγική αυτή. Έχουμε πιο πολλούς στόχους σήμερα στην Ευρώπη από όταν άρχισε να εφαρμόζεται η στρατηγική αυτή. Χάνουμε τον στόχο της απάλυνσης της φτώχειας. Πρέπει να τα πάρουν σοβαρά αυτά οι υπόψη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις χώρες μέλη. Εν τέλει, όταν μιλούμε για την αντιμετώπιση της φτώχειας, η απασχόληση μένει το κύριο φάρμακο. Η δημιουργία θέσεων εργασίας είναι ο καλύτερος τρόπος για να αντιμετωπιστεί η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός. Ακούστηκε όμως μια άποψη στη συζήτηση και στην Ολομέλεια πριν αλλά και στις επιμέρους επιτροπές ότι πρέπει να εξετάσουμε και την ποιότητα της απασχόλησης που δημιουργείται και όλη την υπόθεση του κοινωνικού ντάμπινγκ στην αγορά εργασίας. Όταν εξετάζουμε την ε, στρατηγική Ευρώπη του 2020 πρέπει να επιδιώξουμε απασχόληση ποιότητας που θα έχει ε, θετική επιρροή και στην αντιμετώπιση της ανεργίας. Κάτι πρέπει να προκύψει από τη στρατηγική επενδύσεων. Εδώ υπάρχει και κάποια σύγχυση. Ο ίδιος ο πρόεδρος Γιούνκερ δέχτηκε ότι οι περιφερειακές χώρες της Ευρωζώνης που ε, θεωρούνται υψηλού κινδύνου για τις ιδιώτες επενδυτές θα λάβουν περισσότερες επενδύσεις από το Ταμείο. Όμως τα επενδυτικά έργα θα εξετάζονται από την άποψη της αποδοτικότητας των επενδύσεων. Πρέπει να υπάρξει συντονισμός και ιδίω όταν μιλούμε για τη στρατηγική της Ευρώπης 2020 και για την στρατηγική επενδύσεων. Η Ευρώπη 2020 πρέπει να μπει στην καρδιά των επενδύσεων και τα κριτήρια για την αξιολόγηση των επενδυτικών έργων θα πρέπει να περιλάβουν και μια πραγματική δέσμευση υπέρ των στόχων της Ευρώπης 2020. Και ιδίως όταν μιλούμε για περιφέρειες αυτό οφείλει να γίνει. Ε, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην επενδυτική στρατηγική, μέσα στα πλαίσια της επενδυτικής στρατηγικής δηλαδή, στις ευρωπαϊκές περιφέρειες και ιδίω για την απασχόληση, πραγματική απασχόληση που πρέπει να μπει στην καρδιά της επενδυτικής στρατηγικής για δουλειές δουλειές βιώσιμες και καλής ποιότητας. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Φιγκερέντο από Πορτογαλία. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, κύριοι βουλευτές, ήδη ελεγχθεί ότι η Ευρώπη μπορεί να προχωρήσει αν υπάρχει εμπιστοσύνη. Και αυτό θα επισυμβεί μόνο εάν δεν υπάρχουν αρνητικούς, αρνητικοί παράγοντες. Αυτό που κάνουμε στην Πορτογαλία ήταν να τηρήσουμε τις δεσμεύσεις μας, αλλά θεωρώ ότι η πολιτική απασχόληση δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη ως προς τις δαπάνες, αλλά θα πρέπει να υπάρχει μια καλύτερη κοινωνική δικαιοσύνη έπρεπε στην Πορτογαλία να προβούμε ε, σε πολλές μεταρρυθμίσεις, ιδιαίτερα στον τομέα της εργασίας και όπως ήδη ελέγχθη εδώ στο ημικύκλιο δεν έγινε καμία απόλυση δημοσίων υπαλλήλων. Ήδη έχουμε θετικές ενδείξεις ως προς τον ε, αριθμό των ανέργων, δηλαδή έχουμε μείωση της ανεργίας. Η ανεργία σε μας έφτασε στο 18%. Τώρα έχουμε ένα δίκτυ ανεργίας ε, που είναι πολύ κοντινός με αυτόν του 2011, δηλαδή στην αρχή της διαδικασίας προσαρμογής, όταν ζητήσαμε τη διεθνή αρρωγή. Φυσικά είναι ακόμα υψηλή η ανεργία, όμως έχει μειωθεί. Γιατί δημιουργήθηκαν νέες θέσεις εργασίας. Επίσης, έπρεπε να λάβουμε υπόψη ένα πρόγραμμα κοινωνικής επίγουσας ανάγκης για να μην αφήσουμε κανέναν Πορτογάλο πίσω. Όμως θέλουμε να καταπολύσουμε και τη φτώχεια και να προωθήσουμε τις ε, επενδύσεις. Προσπαθήσαμε να εξισορροπήσουμε την κατάσταση με αποφασιστικότητα και ευθύνη. Η στρατηγική 2020 είναι ύψης της σημασίας και για την Πορτογαλία. Θεωρούμε ότι η Ευρώπη 2020 θα έχει θετικές επιπτώσεις και στην Πορτογαλία για να δώσουμε θετικές απαντήσεις και μετατρέποντας την Πορτογαλία σε μία πιο ανταγωνιστική χώρα. Μιλάμε για τον επιχειρηματικό κόσμο, για την πρόθεσή του, για την απασχόληση και για την ευέλικτη εργασία. Επίσης, αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι η απόκτηση πρώτης εργασίας και η καταπολέμηση των μακροχρονίων ανέργων. Αυτά τα στοιχεία είναι αποφασιστικής σημασίας για να καταπολεμήσουμε μια μεγάλη μάστιγα που είναι η ανεργία των νέων, έτσι ώστε να έχουμε μια Ευρώπη πιο δίκαιη, πιο ανθρώπινη και πιο αλληλέγγυα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Γιάννη Σαράβικ από την Τσεχία. Έχετε το λόγο παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Όπως και προηγούμενοι ομιλητές, έτσι και εγώ θέλω να αναφερθώ στο επενδυτικό πακέτο Juncker. Αυτό που, συζητά, που συζητήσαμε δηλαδή και σήμερα το πρωί και εξακολουθούμε να συζητάμε και τώρα. 315 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό είναι το ποσό. 21 δισεκατομμύρια βέβαια αρχικά που θα πολλαπλασιαστούν επί 15. Αυτή θα είναι η μόχλευση. Είναι αυτό ρεαλιστικό όμως. Είναι εφικτό. Τα σχέδιά μας είναι πολύ φιλόδοξα και όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος. Όταν κοιτάω τις επιπτώσεις των επενδύσεων επί του περιβάλλοντος, διαπιστώνω ότι είμαστε εξίσου φιλόδοξοι. Όταν στηρίζουμε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, επίσης είμαστε φιλόδοξη εξίσου, για όταν θέλουμε να προστατεύσουμε τα δικαιώματα των καταναλωτών, τα ανθρώπινα δικαιώματα κλπ. κλπ. Όλα αυτά όμως μειώνουν την ανταγωνιστικότητά μας σε σχέση με άλλες οικονομίες όπως η κινέζικη. Οι οικονομικές μας πολιτικές βασίζονται ξένιες που έχουν να κάνουν με την μόνιμη ανάπτυξη ή με το γενικό δικαίωμα στην ευημερία. Σήμερα και πρόσφατα ακούμε κάποιες επικίνδυνες απόψεις που αντιβαίνουν μάλιστα σε παλιές παραδόσεις ότι τα χρέη δεν πρέπει να ακολουθήσουν την πορεία που ακολουθούσαν παλιά. Μια που ο Επίτροπος Τάισεν τελικά δεν μπόρεσε να συμμετάσχει σε αυτήν την συνάντηση, μας έχει μείνει χρόνος, μας έχει περισσέψει χρόνος για παρεμβάσεις. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη μέθοδο του Catch the Eye. Υπάρχει κάποιος ακόμα που θέλει να πάρει το λόγο παρακαλώ αρκεί να μας κάνετε ένα νεύμα ότι θέλετε να πάρετε το λόγο, παρακαλώ. Ποιος άλλος θέλει το λόγο. Ελίσα Φερέιρα. Η Ελίζα Φερέιρα. Ευχαριστώ πολύ. Η σημερινή μας συζήτηση είναι πολύ σημαντική. Επίκαιρη. Πρέπει όμως να είμαστε προσεκτικοί με τους όρους που χρησιμοποιούμε. Και το λέω αυτό γιατί κατά τη διάρκεια της κρίσης και μετά από την κρίση χρησιμοποιούμε όρους όπως διορθωτικές μεταρρυθμίσεις ή φιλική προς το περιβάλλον ανάπτυξη ή Ακόμα μιλάμε και για την ε, στρατηγική του 2020, χωρίς να συζητάμε το πραγματικό περιεχόμενο αυτών των ενιών. Αν λοιπόν θέλουμε πραγματικό διάλογο, τότε θα έπρεπε να είναι για μας ξεκάθαρο το τι σημαίνουμε με, τις, με τους όρους αυτούς. Όταν μιλάμε για την στρατηγική 2020, συχνά μιλάμε για ευσεβείς πόθους γιατί οι χώρες οι οποίες χρειάζονται περισσότερα για αυτού του είδους ε, επενδύσεις, για να έχουν ανάπτυξη, για να έχουν σύγκληση, για να βγουν από την κρίση, οι χώρες αυτές δεν έχουν το περιθώριο ε, λιγμών που χρειάζονται δημοσιονομικά για να επενδύσουν ακριβώς πάνω σε αυτά. Και ποιο είναι το αποτέλεσμα? Ότι συνεχίζουμε να μιλάμε για τους στόχους του 2020, για διορθώσεις που θα δώσουν ανάπτυξη. Στην πραγματικότητα όμως δεν αφήνουμε περιθώριο διόρθωσης για τις χώρες που βρίσκονται σε αυτή τη διαδικασία. Ένα λοιπόν από τα θέματα που θα πρέπει να συζητήσουμε και να αντιμετωπίσουμε είναι προσοχή όταν μιλάμε για τις αναχώρα ειδικέ συστάσεις. Όταν η, χώρα, η Επιτροπή συζητάει με τις διάφορες χώρες και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να δούμε ποιο είναι το περιεχόμενο ακριβώς των συστάσεων. Να μην είναι ψευής πόθη, αλλά να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, στα νούμερα. Αν οι χώρες μέλη λοιπόν για να απαλλαγούν από τους κάνουν περικοπές και δεν επενδύουν, αν μειώσουν τις επενδύσεις τους στην ε, έρευνα και τις επιστήμες, στην ενέργεια, αν μειώσουν τις δαπάνες τους για την εκπαίδευση, αν μειώσουν παντού, τότε μπορεί να λέτε ότι θέλουμε στόχους το 2020, αλλά πώς θα πετευθούν. Πρέπει να είμαστε σοβαροί λοιπόν όταν συζητάμε και να είμαστε πολύ προσεκτικοί για την ορολογία που χρησιμοποιούμε και να μην συμφωνούμε με κάτι που τελικά το ερμηνεύουν διαφορετικά οι διάφοροι Αυτό είναι το σχόλιο που θα ήθελα εδώ να καταθέσω για να το συζητήσουμε στο μέλλον. Να ξέρουμε ακριβώς για τι πράγμα μιλάμε και να ξέρουμε ποιο είναι το περιθώριο ελιγμών που αφήνουμε μετά τα προγράμματα στις χώρες για να προβούν σε επενδύσεις. Και όταν μιλάμε για τον επενδυτικό πακέτο Juncker, να ξέρουμε θα ενισχύσουμε τη σύγκληση και υπάρχει και κάποιο στοιχείο που να βοηθάει τις λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες της Ευρώπης να υποφεληθούν από κονδύλια ή επικεντρωνόμαστε σε προγράμματα μόνο που δεν έχουν ιδιαίτερο κίνδυνο και σε χώρες όπου είναι πιο ασφαλείς. Αυτό είναι το σχόλιο που θα ήθελα να καταθέσω εδώ και σας ευχαριστώ πολύ που μου δώσατε την ευκαιρία να το καταθέσω. Ευχαριστούμε. Άλλοι ομιλητές, άλλος κανείς. Α, παρακαλώ, εσείς. Στη θέση 99. Ευχαριστώ πολύ. Από την Τσεχική Δημοκρατία, από το Κοινοβούλιο, θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να απαντήσω σε κάτι το οποίο ελέγχθη πολλές φορές κατά τη διάρκεια της ε, διάσκεψής μας, δηλαδή τη, τη μεγάλη διαφορά μεταξύ πλούσιων και φτωχών, αυτό το χάσμα που υπάρχει. Οι επενδύσεις θα πρέπει να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας, αλλά οπωσδήποτε η εργατική τάξη παραμένει φτωχή. Υπάρχουν πολύ αρνητικά στοιχεία στις ε, οικονομίες μας και εάν θέλουμε, αν θέλει το επενδυτικό πρόγραμμα να προωθήσει την οικονομική ανάπτυξη, τότε ε, δεν θα πρέπει παρά να επιλύσουμε το χάσμα μεταξύ πλουσίων και φτωχών και, εν περιπτώσει, να μην γίνει ακόμα πιο μεγάλο αυτό το χάσμα. Άρα δεν μπορούμε να μιλάμε μόνο για αναπτυξιακή πορεία, αλλά και για ένα επίπεδο ζωής για τους εργαζομένους και δεν είμαι μόνος που αναφέρει κάτι τέτοιο. Το έχουν προαναφέρει πολύ. Έχει μεγάλη σημασία να αρχίσει η ανάπτυξη, αλλά ας αποφύγουμε άλλα ζητήματα δυσίωνα. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση, η μερίδα μας αυτή. Σας ευχαριστώ όλους για τη συνεισφορά σας, λέει η κυρία Ουλσκοκ. Τώρα θα δώσω το λόγο στον κύριο Γκουαλτιέρη, τον πρόεδρο της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων και θα υποβάλει τα καταληκτικά του σχόλια για την σημερινή συζήτηση. Ρομπέρτο, έχεις το λόγο. Ευχαριστώ Μαρίτα. Νομίζω ότι ήταν πολύ επικοδομητική αυτή η πρώτη ημέρα κοινοβουλευτικού διαλόγου. Νομίζω λοιπόν ότι προβήκαμε σε μία μεθοδολογική συζήτηση εδώ και πολύ καιρό γιατί πρέπει να υπάρχει ε, διακοινοβουλευτική διαδικασία, πώς θα λειτουργεί, τι προβάλλει και ούτω καθεξής. Τώρα δώσαμε σε αυτή τη μεθοδολογία περιεχόμενο. Αυτά τα ζητήματα είναι ζωτικής ε, σημασίας για όλους και βεβαίως είναι και αλληλένδετα. Η Ευρώπη 2020, η Στρατηγική 2020, το μέσο για τους νέους και ούτω καθεξής είναι μέσα που προβάλλει η Επιτροπή για το 2015. Θα πρέπει να δούμε κατά πόσο αυτό συμβαδίζει με τους μακροχρόνιους στόχους και κατά πόσο θα πρέπει να αναθεωρήσουμε αυτά τα πλαίσια με βάση τους μακροχρόνιους στόχους ως προς την Ευρώπη 2020. Και τέλος, τα μέσα που χρησιμοποιούμε είναι κατάλληλα είναι τα κατάλληλα για να έχουμε μια αποτελεσματική οικονομική πολιτική για να έχουμε μια οικονομική κυβέρνηση. Τουλάχιστον έτσι παρουσίασε το ζήτημα ο κύριος Γιούνκερ και η Επιτροπή. Αυτά είναι ζωτικά ζητήματα και φυσικά είναι και αλληλένδετα. Φυσικά ποτέ δεν μπορούμε να είμαστε ομόφωνοι για όλα Υπάρχει διάσταση απόψεων, αλλά υπάρχουν ορισμένα γεγονότα και αριθμοί που είναι σαφή. Ο Αντιπρόεδρος Κατάινεν μας παρουσίασε πολλά από αυτά. Δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε σε πολλούς από τους στόχους της στρατηγικής 2020 στον τομέα ενέργειας, ανάπτυξης, μείωσης της φτώχειας και απασχόλησης. Δεν χρειάζεται να υπενθυμίσω αριθμητικά στοιχεία για την ανεργία για το επενδυτικό χάσμα επίσης που, για το οποίο μας μίλησε η Επιτροπή, δηλαδή μιλάμε μείωση επενδύσεων κατά 15% μεταξύ 2007 και 2014. Μιλήσαμε για δίκτυ ανεργίας και το συγκρίναμε με αυτό της Ιαπωνίας και τον είπα. Γνωρίζουμε επίσης και παρακολουθούμε την εξέλιξη του ΑΕΠ μετά την παγκόσμια κρίση. Βλέπουμε ότι συμβαδίζουμε με τις είπα μέχρι το 2011 και μετά υπάρχει μεγάλη απόκληση. Εμείς ζήσαμε μια δεύτερη ύφεση και μερικοί από μας ακολούθησαν αποκλίνουσα πορεία, δηλαδή δεν χρησιμοποιήσαμε τις σωστές πολιτικές η πρόσμιξή τους από το 2011 και μετά. Γι' αυτό υπήρξε και αυτή η διαφοροποίηση και η δεύτερη ύφεση. Δεν μπορέσαμε να αποφασίσουμε ποια στοιχεία αυτής της πρόσμιξης πολιτικών θα θέσουμε σε εφαρμογή αλλά δεν μπορούμε να αρνηθούμε πλέον ότι η έκβαση ήταν κακή δεν ανταποκριθήκαμε στους στόχους, γι' αυτό θα πρέπει να ε, επανεκτιμήσουμε τις πολιτικές μας και την πρόσμιξη αυτή την χρήση πολλών πολιτικών. Αυτό ακριβώς μας είπε και ο Γιούνκερ. Μας είπε ότι δεν θέλει να ε, μιλήσω για διακυβέρνηση. Θέλω να μιλήσω για κυβέρνηση. Εμείς είμαστε μια οικονομική κυβέρνηση και θα πρέπει να προσπαθήσουμε να μειώσουμε τα αρνητικά στοιχεία. Μας το έδωσε με, όλα αυτά με απλά λόγια και μίλησε για μια οικονομική στρατηγική. Εμείς ως κοινοβουλευτικοί θα πρέπει να αναλύσουμε αυτή την πρόταση και να τη σχολιάσουμε κατά την άποψή μου εισαγάγει μία αλλαγή σε σχέση με το παρελθόν. Δηλαδή η απόκληση δεν αρκεί. Έχουμε να κάνουμε με μια Ευρωπαϊκή Επιτροπή που έχει εκλεγεί διαφορετικά από το παρελθόν, η οποία μας ε, παρουσιάζει το περίφημο τρίγωνο αυτή την πολιτική δηλαδή που συνίσταται σε ένα επενδυτικό πρόγραμμα, διότι το επενδυτικό χάσμα ε, είναι κάτι το υπαρκτό και το αναγνωρίσαμε. Επίσης θα πρέπει να επιταχύνουμε τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και θα πρέπει να προωθήσουμε μια δημοσιονομική εξυγίανση που να τάσεται υπέρ της ανάπτυξης. Και υπάρχει και αυτό το κοινωνικό στοιχείο το οποίο αναγνωρίζουμε πλέον. Δηλαδή, κοινωνικό έλλειμμα που υπήρχε μέχρι τώρα. Δεν είχαμε λάβει υπόψη την κοινωνική διάσταση στην οικονομική μας πολιτική. Αυτή είναι μια πολιτική πρόταση την οποία θα πρέπει να αναγνωρίσουμε. Είναι συνεκτική, έχει συνεκτικά στοιχεία που αποτελούν πρόκριμα μίας πολιτικής γραμμής. Θα πρέπει να μπορούμε να συνοψίσουμε την πολιτική μας σε λίγες λέξεις και μπορεί κανείς να συμφωνήσει ή να διαφωνήσει. Άρα οι εξελίξεις είναι θετικές κατά την δική μου άποψη και με βάση αυτά που άκουσα και συζητήσαμε θα ήθελα να σχολιάσω αυτά τα τρία στοιχεία του τριγώνου για να δούμε πώς θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε ώστε η στρατηγική να γίνει πιο αποτελεσματική. Εδώ δεν σχολιάζουμε απλώς, δεν είμαστε παρατηρητές, ούτε δημοσιογράφοι, ούτε οικονομολόγοι. Είμαστε ε, κοινοβουλευτικοί παράγοντες και θα πρέπει να ασκήσουμε το ρόλο μας και τα καθήκοντά μας. Θα πρέπει να πραγματώσουμε αυτή τη στρατηγική, να την κάνουμε όσο πιο συνεκτική γίνεται. Άλλοι βεβαίως μπορεί να προβάλλουν εναλλακτικές στρατηγικές για το, για το εκλογικό μας σώμα στο μέλλον. Τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν για την επιτυχία αυτής της στρατηγικής. Μιλάμε καταρχήν για το επενδυτικό πρόγραμμα. Είναι το πρώτο σημείο του τριγώνου. Δεν θα επεκταθώ γιατί θα το συζητήσουμε αύριο. Υπάρχουν όμως δύο στοιχεία όπου θα πρέπει να προσπαθήσουμε να συνεργαστούμε το Ευρωπαϊκό με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Εμείς θα ε, ορίσουμε τον κανονισμό που ε, προσδιορίζει την εμβέλεια αυτών των ε, ταμείων και γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τη λογοδοσία αυτού του προγράμματος με την Μαρίτα Ούλτσκοκ και με άλλους έτσι ώστε να προσδώσουμε τη σωστή λογοδοσία σε αυτό το πρόγραμμα. Και υπάρχει και το θέμα της γεωγραφικής ε, εξισορρόπησης, γιατί δεν μπορούμε να ορίσουμε το επενδυτικό σχέδιο αναχώρα, όμως θα πρέπει να υπάρχει γεωγραφική ισορροπία. Επίσης, θα πρέπει να δώσουμε έναν πανευρωπαϊκό χαρακτήρα σε αυτό το επενδυτικό πρόγραμμα. Αυτό είναι ένα αντάλλαγμα για να έχουμε μεγαλύτερη συμμετοχή των κρατών μελών στο επενδυτικό σχέδιο και το Ταμείο Επενδύσεων. Και γι' αυτό ακριβώς η Επιτροπή θέλει να ε, εξορροπήσει αυτό το σχέδιο, αλλά θα θέλαμε να πείτε στις κυβερνήσεις σας ότι θα πρέπει να είναι δραστήριες γιατί δεν μιλάμε μόνο για μόχλευση κοινοτικών πόρων, αυτό είναι θέμα της Επιτροπής ε, Προϋπολογισμών, αλλά να σειρεύσει και εθνικό χρήμα. Τη στιγμή που δεν θα συμπεριλαμβάνεται στη διαδικασία ελλημάτων, προσδιορισμού του ελλείμματος. Θα το συζητήσουμε αύριο και θα δούμε κατά πόσο μπορούμε να βελτιώσουμε το πρόγραμμα αυτό. Υπάρχει το δεύτερο στοιχείο, το οποίο είναι και το πιο δύσκολο. Δεν μπορεί να μας βρει σύμφωνους πάντα. Πρόκειται για την δημοσιονομική εξυγίανση και ολοκλήρωση και θα πρέπει να αναγνωρίσουμε το εξής. Εάν ε, δεν είναι φιλική προς την ανάπτυξη, τότε δεν υφίσταται η δημοσιονομική ολοκλήρωση. Άρα είναι ύψη της σημασίας αυτή η πτυχή του ζητήματος και η Ελίζα Φεϊρέρε πολύ σωστά μας μίλησε για το ότι θα πρέπει να προωθήσουμε μία φιλική προς την ανάπτυξη, φορο, ε, δημοσιονομική με συγχωρείτε, ολοκλήρωση. Αυτό το είδαμε και στην ανακοίνωση για την ευελιξία, καλύτερη προσαρμογή στον οικονομικό κύκλο και κατανοούμε ότι υπάρχει ένα ε, πολύ σημαντικό στοιχείο το οποίο θα πρέπει να ληφθεί υπόψη διότι η ευελιξία, ευελιξία σημαίνει ότι δεν αλλάζουμε τους κανόνες, απλώς θα πρέπει να εφαρμόσουμε τους κανόνες καθεαυτούς. Και απαντώντας στο συνάδελφο από τη Bundestag που μίλησε για το ότι δεν θα πρέπει να αθετηθούν οι κανόνες, αλλά και η μη εφαρμογή των κανόνων αποτελεί αθέτηση. Γιατί ε, αν μιλάμε για χρονική απόκληση μεσοπρόθεσμα και δεν εφαρμόσουμε το άρθρο 5 του κανονισμού, το οποίο δεν εφαρμόστηκε ποτέ επί χρόνια, τότε πάλι τι κάνουμε, παραβιάζουμε τον κανόνα, τους κανόνες. Χαιρετίζουμε το γεγονός ότι η Επιτροπή θα εφαρμόσει τους κανόνες πλήρως και δεν θα ξεχάσει ένα μέρος τους. έτσι ώστε να υπάρχει αυτόματη εφαρμογή όλων των μερών, διότι μιλάμε για μια οικονομική κυβέρνηση και όχι διακυβέρνηση όπως είπε ο Γιούνκερ. Άρα τα δύο αυτά στοιχεία και το νέο επενδυτικό, η νέα επενδυτική ρήτρα καθώς και η ρήτρα για την επενδυτική μεταρρύθμιση μας επιτρέπουν την δημοσιονομική εξυγίαση που θα είναι φιλική προς την ανάπτυξη. Πολλοί λένε γιατί δεν εφαρμόζουμε την ρήτρα αυτή έτσι ώστε να υπάρχει ένα σκέλος διορθώσεων από τις, ως προς αποκλήσεις που υπήρξαν σε ορισμένες χώρες. Θα το κάνουμε στο μέλλον, πιστεύω, έτσι ώστε να ενθαρρύνουμε τις παραγωγικές επενδύσεις και να ορίσουμε τον προϋπολογισμό της επόμενης χρήσης. Να γίνει η καλύτερη δυνατή χρήση αυτής της ρήτρα δηλαδή, έτσι ώστε οι εθνικοί προϋπολογισμοί να εστιάσουν την προσοχή τους στις επενδύσεις και να υπάρξει και σωστή δημοσιονομική ευθύνη. Τέλος, ως προς τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, νομίζω ότι με την ανακοίνωση μπορούμε να αποφύγουμε τον κίνδυνο που ε, ζήσαμε μέχρι τώρα, δηλαδή να επιλύσουμε τα ε, σοβαρά προβλήματα και να μιλήσουμε για σύγκληση και, και ένα τρόπο ιδιωτικοποίησης όλων αυτών των δεδομένων. Συμφωνώ με τον Σαραζένο θα πρέπει να δούμε πώς οι συστάσεις που προβάλλονται σε συγκεκριμένες χώρες μπορούν να είναι πιο δεσμευτικές αλλά πιο δημοκρατικές. Ε, λαμβάνοντας υπόψη τον επιμερισμό αρμοδιοτήτων μεταξύ Ευρωπαϊκού και Εθνικών Κοινοβουλίων. Η σωστή, η νομιμότητα μάλλον σημαίνει σύγκληση και συντονισμό οικονομικών πολιτικών που χρειαζόμαστε και την αρχή του ownership γιατί διαφορετικά δεν θα υπάρξουν μεταρρυθμίσεις. Επίσης θα δούμε τι συμπεριλαμβάνεται στις μεταρρυθμίσεις. την ανακοίνωση για την ευελιξία γίνεται λόγος για αυτές τις μεταρρυθμίσεις. Μιλάμε για τον τομέα της απασχόλησης, επενδύσεις για δημιουργία απασχόλησης. Άρα και η συζήτηση για τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις είναι ύψης της σημασίας για το μέλλον. Τέλος, Εν συμπεράσματι, θα ήθελα να πω τα εξής. Υπάρχει μία αιτιώδη συνάφεια μεταξύ αυτών των πολιτικών, δηλαδή η οικονομική πολιτική με τη μακροχρόνια στρατηγική του 2020. Συμφωνώ με πολλές από τις υποδείξεις του γερουσιαστή Γκουεριέρη, ο οποίος μίλησε για το ότι θα πρέπει να συμβαδίσει η οικονομική πολιτική του εξαμήνου με τη στρατηγική 2020. Άρα αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε το περιεχόμενο, την ε, διακυβέρνηση και θα ήταν συνετό η Επιτροπή να αναθεωρήσει τη στρατηγική στο σύνολό της. Διαφορετικά θα επρόκειτο για ένα γραφειοκρατικό εγχείρημα. Τώρα χτίζουμε μία νέα πολιτική και οικονομική στρατηγική. Ελπίζω να μην ε, πνίξουμε τη νέα ανάκαμψη. Θα πρέπει να προωθήσουμε αυτή την στρατηγική και να διαμορφώσουμε εκ νέου τη στρατηγική 2020 με βάση την τρέχουσα, τις τρέχουσες εργασίες. Πολύ καρποφόρα λοιπόν ήταν η συζήτηση. Σας ευχαριστώ όλους για τη συμμετοχή σας και για τη συνεισφορά σας. Σήμερα στις 7 ο Επίτροπος Μοσχοβησή θα βρίσκεται στο ε, δείπνο μας και ο Μάρτιν Σούλς, ο πρόεδρος του Λετωνικού Κοινοβουλίου και δυνάμει του άρθρου 13 θα συνεχίσουμε με τις εργασίες της διάσκεψής μας με στα πλαίσια του διακοινοβουλευτικού διαλόγου και θα εστιάσουμε την προσοχή μας σε άλλα ζητήματα. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε στο δείπνο μας και αύριο για τη δεύτερη μέρα εργασιών. Γεια σας.